Please sit down. We have to go. Please sit down. We have to go. Καθίστε. Πρέπει να μείνουμε στο χρόνο μας, στο βαθμό του δυνατού. Ε, καλωσορίζω βέβαια ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου είναι παρόν και, θα, ε, και θα καλωσορίσει όλους σας, αλλά εγώ καλωσορίζω ε, τον ε, κύριο Μπούζεκ ε, που με την παρουσία του τιμά την έκτακτη συνεδρίασή μας συνδιοργανώνεται η συνεδρίαση αυτή από κοινού με την Υποεπιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα η πρόεδρος Χάουταλα είναι εδώ ε, όπως επίσης ε, και ο πρόεδρος ε, της αντιπροσωπείας με τη Λευκορωσία και τις Εούρονες, δηλαδή συνάδελφοι Βιγένιν και Προτασίεβιτς. Καλωσορίζω και τις άλλες παρούσες προσωπικότητες, τον κύριο Ενατάντησους, ο οποίος είναι υφυπουργός εξωτερικών της Λιθουανίας και εκπρόσωπος ε, της ε, Προεδρίας της ΟΑΣΕ, ο Επίτροπος ε, Φίλε, ο οποίος πρόσφατα πήγε στη Λευκορωσία και μπορεί να μας αναφέρει σχετικά με την αποστολή του, ο πρέσβης Άρενς, ο οποίος είναι και ο πρόεδρος αντιπροσωπείας των παρατηρητών της ΟΑΣΕ και του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών κλπ. Είναι ο, επίσης εδώ ο κύριος Αλεξανδράου που εκπροσωπεί την Ένωση ε, της, ε, των ε, Δημοσιογράφων της Λευκορωσίας που πήρε το γραφείο Σαχάροφ το 2004 όπως επίσης και ο Φραβεσμένος το 2008. Είναι παρόν. Μετά από τις ε, πρόσφατες ε, διαδηλώσεις και την ε, ματοχυσία στην Λευκορωσία μετά από τις προοδρικές εκλογές δεν έχουμε ως στόχο να συζητήσουμε μόνο αυτό το θέμα αλλά είναι ως θέμα σήμερα και η συζήτηση για τις σχέσεις μας με την Λευκορωσία. Αύριο θα συνεδριάσει η διάσκεψη των Προέδρων για να εγκρίνει την αποστολή μιας αντιπροσωπείας μας στη Λευκορωσία. Φυσικά θα εξεταστεί και η απόλυξη της συζήτησής μας σήμερα ούτως ώστε να οριστεί και το πλαίσιο αυτής της αποστολής. Πρέπει να σας πω ότι πριν από, την, αυτήν μας τη συνάντηση ε, συνάντησα τον ε, Υπουργό Εξωτερικών της Λευκορωσίας και εξέφρασα την επιθυμία ε, να μπορέσει η αποστολή μας ε, να ε, έχει και την αιγίδα της λευκορωσικής κυβέρνησης. Είναι πολύ σημαντική η συνάντησή μας σήμερα. Αλλά ε, θα πρέπει να δώσω το λόγο στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, τον οποίο χαιρετίζω και ευχαριστώ για την παρουσία του. Έχετε το λόγο, πρόεδρε Μπούζεκ. Ευχαριστώ, κύριε πρόεδρε. θα πω εκ μιας αρχής ότι ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η μέρα σήμερα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χαίρομαι που είναι παρόντες οι εκπρόσωποι της λευκορωσικής δημοκρατικής αντιπολίτευσης, των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης και της κοινωνίας των πολιτών. Βρίσκονται σήμερα μαζί μας τα πρόσωπα αυτά. Σας δέχθηκα σήμερα το πρωί και συζητήσαμε σε βάθος την κατάσταση αγαπητοί φίλοι, αλλά αυτό δεν αρκεί. Οι συζητήσει μας θα πρέπει να είναι διαφανής για την κατάσταση στην ε, Λευκορωσία, για τα όσα συνέβησαν και για το τι μπορούμε να πράξουμε στο μέλλον ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ζητήσουμε λοιπόν την συμβουλή σας. ώστε να μας πείτε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Ο λαός της Λευκορωσίας είναι καλοδεχούμενος στην ευρωπαϊκή οικογένεια ελεύθερων δημοκρατικών εθνών και σας αναγνωρίζουμε ως εκπροσώπους, των, ως εκπροσώπους της χώρας σας. Πρώτα θα εκφράσω την αλληλεγγύη μας μαζί σας με, με τον λευκορωσικό λαό. Όλοι μας παρακολουθήσαμε προσεκτικά τα γεγονότα στο Μίνσκ και εγώ ήδη από την 20η Δεκεμβρίου ήμουν σε διαρκή επαφή με τον πρόεδρο κύριο Αλμπερτίνη, τον οποίο και ευχαριστώ για την διοργάνωση της παρούσας συνεδρίασης, καθώς επίσης και με την κυρία πρόεδρο Χάουταλα, τον κύριο Γιγένιν, καθώς και τον κύριο Προτασίεβιτς. Ήμασταν λοιπόν σε διαρκή επαφή. Ευχαριστώ ιδιαίτερα και τον Επίτροπο κύριο Φίλερ, με τον οποίο έχω μιλήσει κατ' επανάληψη για να συζητήσω τα διάφορα συναφή θέματα. Ε, παρόν είναι και, παρούσα μάλλον είναι και η Προεδρία του ΟΑΣΕ. Με τις απόψεις που θα εκφράσουμε σήμερα θα δείξουμε ότι στερείται δημοκρατικής νομιμοποίησης η κυβέρνηση Λουκασένκο. Και από αυτή την άποψη είναι απαραίτητο να επανεξεταστεί η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στο Μίνσκ. Κάτι που θα έπρεπε να αρχίσει ήδη από τώρα η επανεξέταση αυτή. Ας αρχίσουμε λοιπόν και ας θεωρήσουμε την παρούσα συνεδρίαση ως αυτό που λέγουν οι αγγλόφωνοι brainstorming, δηλαδή όπου καθένας καταθέτει τις ιδέες του. Πρώτη προτεραιότητα θα πρέπει να είναι να ζητήσουμε από τις αρχές να απολύσουν από τις φυλακές όλους όσοι ακόμη κρατούνται, να εγκαταλείψουν τις βαριές κατηγορίες που έχουν απαγγείλει σε 31 ακτιβιστές και επίσης σημαντικό είναι να προσφερθεί η απαραίτητη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αμέσως σε, ορισμένους, ε, σε ορισμένα μέλη της λευκορωσικής κοινωνίας τα οποία εδάρισαν ανηλιώς. Εύχομαι λοιπόν σε όλες και όλους μια καρποφόρα συνεδρίαση και σας ενθαρρύνω να εκφράσετε τις απόψεις σας σχετικά με το πώ θα πρέπει να προχωρήσει η στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στη Λευκορωσία. Ευχαριστώ και πάλι του φίλου μα από τη Λευκορωσία για την παρουσία του εδώ, η οποία θα επιτρέψει η συζήτησή μα να γίνει και βαθύτερη και πλατύτερη και αναμένουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα από την σημερινή συζήτηση σχετικά με το πώς να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό στο μέλλον. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό ερώτημα που ε, οφείλουμε να θέσουμε όλοι. Σας ευχαριστώ λοιπόν κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ χρήσιμη η τοποθέτησή σας για να μπορέσουμε να οριοθετήσουμε το πλαίσιο της συνάντησής μας. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Μερικές αρχικές πληροφορίες, πρώτη τεχνικού χαρακτήρα. Τα λευκορωσικά ε, η λευκορωσική διερμηνία ακούγεται από το κανάλι 17 αν οι φιλοξενούμενοι μας θέλουν να ακούσουν ε, τη συζήτηση στη γλώσσα τους. Εγώ προβλέπω τα εξή ω διαδικασία σήμερα. Πρώτο τμήμα της συζήτησης αφορά στην εκλογική διαδικασία, στην μετεκλογική κατάσταση. Ο πρεσβής κ. Άρεντς θα μας μιλήσει για αυτό το σενάριο. Μετά θα μιλήσουν οι δύο νικητές του βραβείου Ζαχάροφ, ο κύριος Μιλικίεβιτς και ο κύριος Αλεξάνδροφ, που θα μας περιγράψουν την κατάσταση στη χώρα. Και για το δεύτερο τμήμα, σχετικά με τη θέση της διεθνούς κοινότητας, θα μιλήσουν ο Επίτροπος, ο κύριος Φίλε και ο Λιθουανός Υφυπουργό υφυπουργός εξωτερικών ο οποίος θα μας αναφέρει πως έχει κατάσταση στην ΟΑΣΕ. Παρακαλώ τους ομιλητές να είναι σύντομοι, να μιλήσουν πέντε λεπτά ο καθένας, ούτω ώστε να έχουν στη συνέχεια την δυνατότητα να απαντήσουν στις ερωτήσεις των συναδέλφων. Προβλέπετε Επίσης και η τοποθέτηση της κυρίας Νίκολάιεβα η οποία θα μιλήσει στη συνέχεια. Κύριε Πρεσβευτά, κύριε Άρενς. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ ήμουν επικεφαλής της αποστολής παρακολούθησης μακροχρόνιας στην ε, Λευκορωσία από το 2006 στο 2008 και 2008-2010 εξ ονόματος της ΟΣΑ και του Γραφείου για τους Δημοκρατικούς Θεσμούς και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Όλες αυτές οι αξιολογήσεις μας ήταν αρνητικές. Υπήρξαν κάποιες βελτιώσεις σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές. Αλλά δεν έχει αντιμετωπιστεί μια χωρία πολύ σημαντικών θεμάτων και τα πραγματικά σημαντικά θέματα είναι καταρχήν το άκαμπτο του πολιτικού συστήματος στη Λευκορωσία και επίση ο τρόπο με τον οποίο γίνεται η καταμέτρηση των ψήφων και η πρώιμη διαδικασία ψηφοφορία Το 2010 συναντήθηκα όλου του υποψηφίου που ήταν αντίπαλοι του κυρίου Λουκασέγκο και μου είπαν ότι κανεί του δεν έχει εμπιστοσύνη στην εκλογική διαδικασία. Ενώ οι επίσημοι συνομιλητέ τονίζουν ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε αυτή τη φορά την πρόοδο που επετελέστη στην ε, Λευκορωσία. Ένας υποψήφιος είπε κάτι το οποίο θέλω να το τονίσω γιατί είναι πολύ σημαντικό. Είπε ότι έχουμε ένα, μια στρατιωτική μονάδα που κάνει γυμναστικές ασκήσεις. Κάποιος πηγαίνει, προσπαθεί να σηκωθεί από να κάνει έλξη σε μία μπάρα και δεν τα καταφέρνει, αλλά μετά συνεχίζει, φεύγει και του λένε 5 στα 5 εξαιρετική απόδοση. Αυτό το ίδιο πράγμα γίνεται και στην περίπτωση των εκλογών. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να καταλάβουμε τι είναι σημαντικό και τι είναι επουσιώδες σε αυτές τις περίφημες βελτιώσεις που έλαβαν χώρα στην Λευκορωσία. Έχουμε εντοπίσει πολλά αρνητικά σημεία, αλλά αυτά μπορείτε να τα δείτε στο έγγραφό μας, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω και γι' αυτό θα σταθώ μονάχα στα πολύ σημαντικά θέματα. Στην αρχή της αποστολής μας, ο επικεφαλής της, της του Προεδρικού Γραμμίου, ο κύριος Μακέι μου είπε ότι περίμενε μια θετική αξιολόγηση από την πλευρά του, της ΟΑΣΕ και το ίδιο μου είπε και ο Υπουργό Εξωτερικών. Είπαν ότι έχουν επέλθει πραγματικές βελτιώσεις και δεν μπορούσαν να επιτύχουν τίποτα περισσότερα από όλα αυτά. Οι οποιασδήποτε μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να γίνουν σταδιακά. Εγώ νομίζω ότι αν εξασφαλιστεί πραγματικά να γίνει σωστά η καταμέτρηση των ψήφων, αυτό θα ήταν πολύ σημαντικό. Αλλά οι δύο εκλογές που παρακολούθησα ουσιαστικά ξεκινούσαν σε πολύ νωρίς πρωινέ ώρες και τελείωναν πολύ νωρίς μέσα στο μεσημέρι, το οποίο δεν βοηθούσε τη διαδικασία. Τώρα, το θέμα της ε, αξιολόγηση των εκλογών το, η εκλογική επιτροπή ταυτίζεται με το κράτος, το κράτος ταυτίζεται με τον πρόεδρο και ο πρόεδρος ταυτίζεται τον εαυτό του με το λαό. Αυτό είναι και το μήνυμα του συνεδρίου όλων των Λευκορώσων που είναι αυτοί που υποστηρίζουν τον πρόεδρο και οι οποίοι παρουσιάζουν τους πολίτες της χώρας αυτής ως ευτυχείς και ικανοποιημένους. Και αυτό ανταρακτώνεται και στα μέσα ενημέρωσης. Εγώ μίλησα με πάρα πολλούς στη Λευκορωσία και πολλοί από αυτού είπαν ότι είναι πιο ικανοποιημένοι που ζουν σήμερα στο Μίνσκ από την εποχή που επί Σοβιετική Αυτοκρατο... Ε, ζούσαν στη Μόσχα. Αλλά είναι απόλυτα ανεπαρκή και υπανάπτυκτου χαρακτήρα κατά κάποιο τρόπο τα κόμματα τη αντιπολίτευση, μερικά από τα οποία δεν έχουν ακόμα γίνει δεκτά για να καταγραφούν ω επίσημα κόμματα. Πολλέ φορέ υπάρχει εντύπωση ότι τα μέλη της ε, εκλογικής ε, επιτροπής που προσδιορίζονται από κόμματα της αντιπολίτευσης είναι ξενόφερτοι και πράκτορες ξένων συμφερόντων και πρέπει να τους κρατάμε στην άκρη. Οι πιο σημαντικές θέσεις βρίσκονται πάντα στα χέρια του κυβερνώντος κόμματος ή σε οργανισμούς που πρόσκυνται στις κυβερνητικές δυνάμεις. Υπάρχει λοιπόν ένας φαύλος κύκλος. <clears throat> Αν ο κύριος Σάνικοφ ο οποίος είναι ο επικρατέστερος εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης παίρνει μονάχα 2,5% στις εκλογές, γιατί να εκπροσωπούνται τα κόμματα της αντιπολίτευσης στις εκλογικές επιτροπές. Επομένως είναι πραγματικά μεγάλα τα προβλήματα. Μετά από την εμπειρία που είχαμε για την διεξαγωγή της εκλογικής εξαρτίας, πρέπει να πω ότι έχουν γίνει δύο σφάλματα. Καταρχήν υπήρξε έλλειψη Ενότητο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εννέα υποψήφοι που είναι κυρίως άγνωστοι δεν βοηθούν τα πράγματα. Δεύτερον, δεν υπήρξε επαγγελματικός χαρακτήρας κατά τη διάρκεια των εκλογών. Ο στόχος δεν ήταν να πούν στον κόσμο που ήξερε αυτά που ήθελαν να ακούσουν, αλλά να μπορέσουν να ανατρέψουν την κατάσταση και να πάρουν εξουσία από τον κύριο Λουκασέγκο. Η τελευταία μου παρατήρηση τώρα είναι το θέμα του ρωσικού ρόλου στις εκλογές αυτές πριν από τις εκλογές, ο πρόεδρος Μετβέντιεφ επέκρινε τον πρόεδρο Λουκασέγκο. Και αυτό οδήγησε ορισμένου να περιμένουν ότι θα άλλαζαν τα πράγματα και θα υπήρχε μια διαφορετική στάση από τη Ρωσία για τα θέματα αυτά. Επειδή οι, οι κακές σχέσεις με τη Ρωσία δεν υποστηρίζονται από το λαό και πολλοί, πολλοί υποψήφοι της αντιπολίτευσης υποστήριξαν το ότι φταίει ο Λουκασέγκο για τις ε, καλές, για τις κακές αυτές σχέσεις. Αλλά στη συνέχεια αναφέρθηκε ότι είναι πολύ καλές οι σχέσεις των δύο πλευρών. Τουλάχιστον σε μία περίπτωση έγινε σαφές ότι η αξιολόγηση από, τους, ε, από τις χώρες της ε, Ομοσπονδίας Πλώην Σοβιετικών Κρατών έχουν μια ριζικά διαφορετική αντιμετώπιση από αυτή του ΟΑΣΕ. Η κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία της ΟΑΣΕ με τον κ. Τόνι Λάου επικεφαλής ήταν εξαιρετικά καλή στο έργο της και θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου γι' αυτό γιατί υπήρξαν πολλές δυσκολίες στο παρελθόν σε σχέση με την Προεδρία της ΟΑΣΕ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Eh, Ευχαριστώ κύριε Πρεσβευτά. Ο κύριος Μιλινκίεβιτς, πρόεδρος του Κινήματος ε, για την Ελευθερία και νικητής του βραβείου Ζαχάροφ του 2006. Μετά θα μιλήσει και η Εύα Νεκλάγεβα, κόρη του Βλαδιμίρ Νεκλάγεβ, ε, υποψήφιου των προεδρικών στις προεδρικές εκλογές και τώρα στη φυλακή. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η λευκορωσική αντιπροσωπεία θεωρεί ότι οι εκλογές ήταν νοθευμένες. Κατά τη γνώμη μας θα πρέπει τουλάχιστον να γίνει ένας δεύτερος γύρος. Συγγνώμη. Οι διερμηνείς μόλις μου ανακοίνωσαν ότι υπάρχει ένα... Ότι μόλις υπάρχει ένα πρόβλημα με την ε, διερμηνία λόγω παρασύτων ε, στην καμπίνα. Παρακαλώ οι διερμηνείς να με ενημερώσουν όταν έχει λυθεί το θέμα των ε, παρασύτων. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να διακόψουμε για μερικά λεπτά για να λυθεί το τεχνικό πρόβλημα. Ένας τεχνικός διορθώνει μόλις τα πράγματα και ελπίζω ότι θα λυθεί σύντομα το πρόβλημα. okay. Μόλις μου είπαν ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε και πάλι. Σας παρακαλώ λοιπόν. Ξαναρχίζουμε παρακαλώ. Κύριε Μιλίνκεβιτς, ζητώ συγγνώμη. Θα επαναλάβω κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν μεταφράστηκα καλά πριν, η δημοκρατική αντιπολίτευση της Λευκορωσίας θεωρεί τις εκλογές αυτές ως νοθευμένες και άδικες. Είμαστε βέβαιοι ότι στην πραγματικότητα ο Λουκασένκο δεν έφτασε το 50% των ψήφων και το λιγότερο που θα έπρεπε να γίνει θα ήταν ένας δεύτερος γύρος εκλογών προ για το καθεστώς ήταν σημαντικό να διαθέτει την ομοποίηση μέσα στη Λευκορωσία και για τις διαβουλεύσεις με την Δύση και με τη Ρωσία η οποία υποστήριζε την, τον Λουκασένκο και τον υποστηρίζει σε όλα τα θέματα. Τούτη τη φορά όμως τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Υπήρχε η ανάγκη να νομοποιηθούν απέναντι στην Δύση ώστε να βελτιώσουν τις σχέσεις κυρίως στην οικονομική σφαίρα. Ταυτόχρονα επιδεινώθηκαν οι σχέσεις με τη Ρωσία. Στην αρχή των εκλογών υπήρχε λοιπόν μια δημοκρατική ατμόσφαιρα. Αλλά στο τέλος, γιατί έγιναν αυτά τα αντίπεινα, γιατί υπήρξε αυτή η αντίδραση των αρχών, γιατί εδάρισαν αθώοι άνθρωποι που συμμετείχαν σε ειρηνικές διαδηλώσεις και γιατί οι αρχές κίνησαν ποινικέ διώξεις κατά 31 ε, ηγετών της αντιπολίτευσης δημοσιογράφων κλπ. Διότι οι αρχές κατανόησαν ότι δεν την χάνουν της υποστήριξης του λαού και γιατί οι διαμαρτυρίες έχουν ενταθεί. Δεν ήταν ορθή η αντίδραση αυτή. Αυτά χρησιμοποιήθηκαν ως προφάσεις. Η αντιπολίτευση δεν είχε σχεδιάσει τέτοιου είδους ενέργειες. Τι θα έπρεπε να κάνει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αντίδραση πρέπει να είναι ξεκάθαρη, συνεπής και να χρησιμοποιηθούν όλες οι οδοί άσκησης πίεσης οικονομικής, διπλωματικής και το πιο σημαντικό θα είναι η άνευ όρον απόλυση των πολιτικών κρατουμένων και αυτών που αντιμετωπίζουν τώρα ποινικέ διώξει. Ο Νίκολα Αυτεχόβιτ και αυτός δεν πρέπει να λησμονηθεί, πολιτικός κρατούμενος. Είναι σημαντικό η Ευρωβουλή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δράσουν ταυτόχρονα. Και οι δηλώσει είναι σημαντικέ, αλλά και οι ενέργειε είναι σημαντικέ από πλευρά των ευρωπαϊκών θεσμών. Πιστεύω ότι αυτές οι πιέσεις ωστόσο δεν πρέπει να οδηγήσουν σε απομόνωση της χώρας μας. Διότι στη χώρα μας, εκτός από αυτούς που υπηρετούν το καθεστώς, υπάρχουν άλλα 9,5 εκατομμύρια Λευκορώσων που είμαστε Ευρωπαίοι. Και δεν θέλουμε να μας σταματήσει κανένα στον δρόμο μας επιστροφή στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Η άποψή μου λοιπόν είναι ότι πρέπει να υιοθετηθεί μια πολιτική σε δύο επίπεδα. Μια, ένα επίπεδο θα είναι οι σχέσεις με το καθεστώς και το άλλο επίπεδο θα πρέπει να είναι οι σχέσεις με την λευκορωσική κοινωνία. Εφόσον οι αρχές απομονώνονται λόγω της πολιτικής τους, παρόλα αυτά θα πρέπει οι πόρτες να μείνουν ανοιχτές για τους λευκορώσους προς την Ευρώπη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν με ρωτήσετε ποιες θα είναι οι πιο αποτελεσματικές κυρώσεις, θα σας πω ειλικρινά ότι οι πιο αποτελεσματικές κυρώσεις κατά πολιταρχικών καθεστώτων είναι η υποστήριξη, ευρεία υποστήριξη στα, μέσα, στα ανεξάρτητα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στην κοινωνία των πολιτών. Θα πρέπει να επανεξεταστεί η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στη Λευκορωσία. Να ιδρυθούν ειδικοί μηχανισμοί που να μας επιτρέψουν να προωθήσουμε τον εκδημοκρατισμό της κοινωνίας Είναι άλλη η ιστορία του διαλόγου με τον Λουκασένκο. Αυτά που έγιναν όμως με τρία χρόνια διαλόγου ήταν σημαντικά επιτεύγματα. Διότι ήδη οι μισοί Λευκορώσοι σήμερα είναι αισιόδοξοι σχετικά με την ευρωπαϊκή πορεία. Θέλουν να επανέλθουν στην Ευρώπη. Αυτό δεν ήταν έτσι στο παρελθόν. Έχουν διπλασιαστεί οι αριθμοί αυτοί. Μόνο 10% Λευκορώσων θα ήθελαν να επιστρέψουν στην ε, Ρώσικη Κοινοπολιτεία, ενώ στην Ουκρανία είναι διπλάσιος ο αριθμός αυτός. Η παραπέρα πορεία των ευρωπαϊκών αξιών είναι σημαντική. Είναι σημαντικό να μιλήσει η Ευρώπη με μία φωνή για την κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στη χώρα μου και οι διάφορες ευρωπαϊκές χώρες να μιλήσουν με μία φωνή. Δεν είναι δυνατόν ορισμένοι να λένε ότι παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και άλλοι να κάνουν ότι δεν βλέπουν τίποτα. Πιστεύω ότι μπορούμε να επιτύχουμε θετικά αποτελέσματα με καλό συντονισμό των ενεργειών μας στην δημοκρατική μας κοινωνία αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι το πιο σημαντικό μας εταίρος. Ο Λουκασένκο θα βγει στην τηλεόραση να πει ότι α, οι Ευρωπαίοι δεν μας θέλουν, είναι κατά της ανεξαρτησίας μας. Πρέπει να καταστήσετε σαφές ότι δεν θέλετε να υποθείτε το καθεστώς, αλλά τους ελεύθερους λευκορώσους. Θα ζητήσω λοιπόν αυτά να υλοποιηθούν. Εκτός από το ψήφισμα λοιπόν πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα. Ελπίζω οι συνάδελφοί μου που συμμετέχουν εδώ να με υποστηρίξουν. Σας ευχαριστούμε για αυτή την ακρόαση που είναι πάρα πολύ σημαντική για μας και κυρίως και για αυτούς που βρίσκονται στις φυλακές. Ε, Ευχαριστώ κύριε Μελίνκεβιτς. Για πέντε λεπτά έχει το λόγο η κυρία Εύα Νεκλάγεβα. Uh, Καλημέρα σας, λέγομαι Εύα Νεκλάγεβα και η θέση μου δεν είναι εδώ. Αντί να βρίσκομαι εγώ σήμερα θα πρέπει ο πατέρας μου Βλαντίβιρ Νεγκλάιεφ με άλλους λαμπρούς και θαραλέους ηγέτες της αντιπολίτευσης στην Πελαρούς θα έπρεπε να βρίσκονται εδώ. Και είναι αυτή η αντιπολίτευση που κέρδισε τις εκλογές. Αλλά στην φρικτή κατάσταση που αντιμετωπίζουμε σήμερα οι νικητές των εκλογών δεν μπορούν να αναγνωριστούν και να είναι εδώ ενώπιόν μας. Αντίθετα λοιπόν από αυτό το οποίο θα πρέπει να συμβεί εδάρισαν ανηλαιώς, ρίχτηκαν στη φυλακή και τώρα αντιμετωπίζουν κατηγορίες που μπορούν να τους κρατήσουν για χρόνια στη φυλακή. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία αυτή να λάβω το λόγο ενώπιό σας και να δώσω φωνή σε όλους τους ε, κρατουμένους συνείδησης και τους οικείους τους, όλους αυτούς που βρίσκονται τώρα στη φυλακή στη Λευκορωσία και χρειάζεται να κατανοήσετε το πόσο κατεπίγουσα είναι η κατάσταση στη Λευκορωσία γιατί έχουμε άτομα τα οποία έχουν ξυλοκοπηθεί ε, πολύ σοβαρά και δεν έχουν ιατρική περίθαλψη. Δεν ξέρουμε σε ποια είναι η, κατάστασή του. Ο πατέρας μου είχε μια μεγάλη ε, κρίση υγείας στην φυλακή το Δεκέμβριο και έκτοτε δεν ξέρουμε καθόλου τι συμβαίνει με αυτόν, τι πιέσεις υφίσταται, αν έχει κάποια ιατρική περίθαλψη και βοήθεια ή όχι. Δεν ξέρουμε τίποτα για όλα αυτά. Και το ίδιο ισχύει και για πολλούς άλλους υποψηφίους, ακτιβιστές, δημοσιογράφους, αγωνιστές των ανθρωπινών δικαιωμάτων που υφίστανται τρομερές πιέσεις. Παραδείγματος χάρη γνωρίζετε ότι ο, ο γιος του Σάνικοφ και της Εντίνα Χαλίπ που είναι τριών ετών ε, απειλούν οι αρχές να τον αποσπάσουν από τους ε, παπούδες του. Και αυτό είναι και βίαιο και απάνθρωπο. Είναι άσκηση τρομοκρατίας η οποία λαμβάνει η χώρα στη Λευκορωσία. Υπάρχει και τεράστια πίεση επίσης που ασκείται σε δημοσιογράφους και ακτιβιστές ανθρωπινών δικαιωμάτων. Μας λένε ότι κάθε μέρα γίνονται νέες συλλήψεις, γίνονται έρευνες στα σπίτια, έρευνες στα γραφεία τους, τους καλούν για ανάκριση από τις μυστικές υπηρεσίες όπου ασκείται και σωματική βία εναντίον τους. Συνεχίζεται λοιπόν η κατάσταση όπως ήταν και στο παρελθόν, επιδεινώνεται μάλιστα και φοβόμαστε πάρα πολύ για τα άτομα που είναι στη φυλακή και δεν απολαμβάνουν ούτε των στοιχειωδών δικαιωμάτων. Θέλω να πω επίσης <clears throat> ότι συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Μιλίνκεβιτς για την ανάγκη να υποστηρίξετε την κοινωνία των πολιτών στη Λευκορωσία αλλά αυτό δεν θα βοηθήσει από μόνο του για την απελευθέρωση όλων των κρατουμένων οι οποίοι πρέπει αμέσως να ελευθερωθούν από τις φυλακές. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένες δράσεις, χρειαζόμαστε στεναρές ενέργειες από τη δική σας πλευρά. Χρειάζεται να κατανοήσετε ότι εσείς έχετε το κλειδί το οποίο θα βγάλει τον πατέρα μου από τη φυλακή και όλους τους άλλους κρατουμένους. Από εσά εξαρτάται το αν όλοι αυτοί οι αγωνιστές της δημοκρατίας θα απελευθερωθούν γιατί βασιζόμαστε πάνω απ' όλα στη διεθνή αλληλεγγύη. Για όλους τους κρατούμενους συνείδηση στη Λευκορωσία και θα περνάνε σαφής η επιλογή σας. Έχετε μονάχα δύο επιλογές. Μπορείτε να κάνετε ένα ψήφισμα να εκδώσετε ένα ψήφισμα το οποίο θα ασκήσει ουσιαστική πολιτική πίεση στη Λευκορωσία και να δώσετε προτεραιότητα σε μια τέτοια στάση έναντι της Realpolitik. Θα πρέπει να τονίσουμε τη σημασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών ελευθεριών που θα πρέπει να υπερισχύσει οικονομικών συμφερόντων. Μόνο έτσι θα μπορέσετε να σώσετε τον κόσμο από τη Λευκορωσία. Ή αλλιώ μπορείτε να ακολουθήσετε μία άλλη οδό η οποία ουσιαστικά θα αποτυπωθεί σε ένα ψήφισμα που θα πείτε κάτι χλιαρό το οποίο θα σημαίνει ότι δεν σας νοιάζει τελικά. Το επίπεδο βίας, το επίπεδο απάνθρωπης αντιμετώπισης από τις αρχές της Λευκορωσίας έχει φτάσει πια μια κορύφωση. Δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτά τα οποία συνέβαιναν πριν από πέντε χρόνια. Θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν μια τελείως διαφορετική αντιμετώπιση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια τελείως διαφορετική και πρέπουσα αντίδραση σε όλα αυτά τα γεγονότα. Σας ευχαριστώ πολύ και πρέπει να πω ότι και σαν κόρη ενός αγωνιστή της ε, δημοκρατίας στη Λευκορωσία πιστεύω και στις συμβολικές δράσεις και φέραμε ε, φουλάρια με τα χρώματα της εθνικής μας σημείας, σημαίας που είναι κόκκινα και λευκά και θα σας τα μοιράσουμε για να διαδηλώσετε και εσείς την αλληλεγγύη σας με αυτόν τον απλό και συμβολικό τρόπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Νικολάγεβα. Δίνω το λόγο στον κύριο Αλεξανδρόφ, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών της Λευκορωσίας, που νίκησε και το βραβείο Ζαχάροφ του 2008. Σας ευχαριστώ και πρώτα θα εκφράσω την ευγνωμοσύνη μας στην Ευρωβουλή για την διαρκή παρακολούθηση της κατάστασης στην χώρα μου. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον πρέσβη κύριο Άρενς και την αποστολή του για την θαυμάσια δουλειά που έκαναν στη Λευκορωσία. Θα ήθελα, θα ήθελα να προσθέσω κάτι ακόμη σχετικά με τις εκλογές που διεξήχθησαν στη χώρα μου. Στην διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας το θέμα της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης έλαβε κυρίαρχο ρόλο, διότι τα μαζικά μέσα ενημέρωσης αποτελούν πλατφόρμα για την δημόσια συζήτηση που περί αυτού πρόκειται εν τέλει στις εκλογές. Εάν δεν υπάρχει ελευθερία του τύπου, εάν υπάρχει περιορισμό στην ελευθερία έκφρασης, εάν δεν υπάρχει η δυνατότητα να γίνει αυτή ανοιχτή δημόσια συζήτηση, δεν μπορεί κανείς να μιλεί για ε, ελεύθερες εκλογές, όσες, όσους καλοπισμούς και αν έκαναν στις διαδικασίες οι αρχές. Ως εκπρόσωπος της κοινότητας των δημοσιογράφων των ελεύθερων μέσων στην Λευκορωσία, θα σας πω ότι ακόμα και πριν από τις εκλογές, στην διάρκεια με τις περιόδους εκείνης που εντός εισαγωγικών ε, την είπαν απελευθέρωση δεν λύθηκαν σημαντικά προβλήματα των μέσων ενημέρωσης. Εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε διοικητική πίεση, οικονομικές διακρίσεις και σημαντικά προβλήματα. Και ξεκάθαρη διάκριση σε βάρος μας. Το πρόβλημα της πρόσβασης στις πληροφορίες είναι σημαντικό και κρίσιμο η σχετική νομοθεσία δεν συμμορφούνται με τις διεθνείς προδιαγραφές. Οι αρχές της χώρας καθαρά, δείχνουν καθαρά την πρόθεσή τους να ρυθμίζουν τα, του διαδικτύου και μάλιστα ιδιαίτερα στις 19 Δεκεμβρίου όταν οι περισσότερες δημοφιλείς ιστοσελίδες του, του διαδικτύου μπλοκαρίστηκαν στη χώρα σε μια προσπάθεια των αρχών να στερήσει από τους πολίτες τις ε, αληθείς πληροφορίες σχετικά με το τι έγινε στην πλατεία ανεξαρτησίας. Σήμερα αντιμετωπίζουμε βαριά, βαριά καταπίεση. Ο μηχανισμός εξακολουθεί να λειτουργεί, ο μηχανισμός καταπίεσης. Δεν σταμάτησε να λειτουργεί στις 19 και 20 Δεκεμβρίου όταν έγιναν πολλές κρατήσεις και πολλοί συμπατριώτες μου κρατήθηκαν διοικητικά. έρευνες, ανακρίσεις ε, ανεξάρτητων δημοσιογράφων συνεχίζονται καθημερινά και τον σύνδεσμο δημοσιογράφων ο επικεφαλής μας σήμερα ανακρίνεται από την ΚΑΚΕΜΠΕ ως μάρτυρας σε μια ε, ποινική δίωξη εναντίον ε, συναδέλφων μας. Η ανεξάρτητη δημοσιογραφία και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών αναμένουν να επιδεινωθεί η κατάσταση. Η καταπίεση σε βάρος των ανεξάρτητων δημοσιογράφων και μέσων θα συνε... και της ε, κοινωνίας των πολιτών θα συνεχιστεί. Μιλώ σήμερα ενώπιον σας όχι μόνο για λογαριασμό του Εθνικού Συνδέσμου ε, Λευκορώσων Δημοσιογράφων αλλά και για να μεταφέρω τις απόψεις ενώ μιας ομάδας ε, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που έχουν συνδυάσει τις προσπάθειές τους σε μια εθνική πλατφόρμα ε, της ε, ανατολικής γειτονίας. Έχουμε λοιπόν μια κοινή δήλωση την οποία έχω εδώ και ε, επιτρέψτε μου να σας αναγνώσω ορισμένα επιμέρους που συναποτελούν το μήνυμά μας προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και την Ευρωβουλή και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφού πρώτα συμφωνήσω με τον κύριο Μίλαν Κίεβιτς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μιλήσει με μια φωνή και να έχει μια συγκεκριμένη θέση ενία απέναντι στην κατάσταση στη Λευκορωσία. Οι οργανώσεις λοιπόν κοινωνίας των πολιτών της Λευκορωσίας ζητούν από τις κυβερνήσεις των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τα θεσμικά της όργανα Ευρωκοινοβούλιο, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Συμβούλιο Υπουργών να κάνουν κάθε τι το δυνατόν για να επιτύχουν την απόλυση από τις φυλακές όλων των κρατουμένων. Αυτό είναι πραγματικά κρίσιμο, κρίσιμη σημασία. Και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να είναι ο πιο αμεσοπρόθεσμος στόχος που πρέπει να έχουμε. Ζητούμε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να μην επιτρέψουν την συμμετοχή των λευκορωσικών αρχών σε προγράμματα της ε, ε, πολιτικής γειτονίας προς Ανατολάς. Καμία συνεργασία μέχρι ότου απολυθούν όλοι οι κρατούμενοι και μέχρι ότου αποσυρθούν οι ποινικέ κατηγορίες. Σας απευθύνουμε έκπληση επίσης να δημιουργήσετε Διεθνή Επιτροπή για την αντικειμενική εξέταση των γεγονότων της 19ης και 20ης Δεκεμβρίου στο Μίνσκ. Σας ζητούμε επίσης να έρθετε σε επαφή με τις λευκορωσικές αρχές, τα αρμόδια υπουργεία, για να σταματήσει η αποπομπή ε, φοιτητών από τα πανεπιστήμια, καθώς και η απόλυση καθηγητών από τα πανεπιστήμια, μόνο επειδή συμμετείχαν σε ειρηνικές διαδηλώσεις. Να συνεχίσετε τις ε, τακτικές επαφές με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στη Λευκορωσία να μειώσετε το κόστος των προξενικών θεωρήσεων για Λευκορώσους πολίτες. Το βασικό μας μήνυμα είναι ότι δεν θα θέλαμε να απομονωθεί η χώρα μας. αλλά θα πρέπει να ληφθούν αυστηρά μέτρα κατά εκείνων που ευθύνονται για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν. Αυστηρά μέτρα και αυστηρή στάση απέναντι στις λευκορωσικές αρχές. Όχι όμως απέναντι στους απλούς πολίτες της Λευκορωσίας, όχι απέναντι στην κοινωνία των πολιτών. Σας ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ κύριε Αλεξανδράου. Ο Λιθανός Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Ινατιαντίτσους, ο οποίος εκπροσωπεί και την Προεδρία της ΟΑΣΕ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ιδιαίτερα τον κύριο Γέρζι Μπούζεκ, τον πρώτο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για αυτή τη συνεδρίαση που αφορά την κατάσταση στη Λευκορωσία. Τα γεγονότα της 19ης και της 20ης ε, Δεκεμβρίου οδήγησαν σε άμεση αντίδραση στην ε, Λιθουανία. Έγινε συζήτηση στο Κοινοβούλιο μας, <clears throat> μια δήλωση για τα θέματα αυτά και την 1η Ιανουαρίου η Λιθουανία ανέλαβε την Προεδρία της ΟΑΣΕ και ο Υπουργός μου, κ. Σασούμπαλης, ε, λαμβάνει μέρος στην διαδικασία ανάληψη καθηκόντων. Ενώ συγχρόνω είναι φανερό ότι η κατάσταση στη Λευκορωσία θα είναι και αντικείμενο συζήτηση στην Βιέννη. Είναι θετική λοιπόν αυτή η ύπαρξη παραλλήλων διαδικασιών και γνωρίζετε ποιε είναι οι αξιολογήσει μα για τι ε, εκλογέ. Δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω αυτά τα στοιχεία. Απλώς θέλω να ξεκινήσω από το γεγονός ότι υπήρξε μια μεγάλη καταστολή της κοινωνίας των πολιτών μετά από τις εκλογές και, ακολούθησε με την ε, απόφαση της κυβέρνησης Λευκορωσίας στις 31 Δεκεμβρίου 2010 να μην παρατείνει την ε, παρουσία της αντιπροσωπείας της ΟΑΣΕ στη Λευκορωσία. Και αυτό καταδεικνύει το πώς καταραίουν οι αρχές της δημοκρατίας, το κράτος δικαίου και οι πολιτικές ελευθερίες στη Λευκορωσία. Να σας δώσω ορισμένα στοιχεία για τις πρόσφατες εξελίξεις στη Λευκορωσία και για τις σχέσεις Λευκορωσίας και ΟΑΣΕ. Ο υπουργό μου ήρθε σε επαφή με τον κύριο Ματίνοφ, τον Υπουργό Εξωτερικών της ε, Λευκορωσίας στις 30 Δεκεμβρίου, προσπαθώντας να αναστρέψει την απόφαση για το κλείσιμο του γραφείου της ΟΑΣΕ στο Μίνσκ, αλλά αυτό δεν καρποφόρησε. Και εγώ επίσης συζήτησα με τον ομολόγο μου, με τον ομόλογό μου την προηγούμενη εβδομάδα. Η απάντηση όμως είναι ότι είναι μια ηλυμένη απόφαση η οποία δεν μπορεί <clears throat> να τροποποιηθεί. Η Λιθουανία ως, προεδρεύουσα της ΟΑΣΕ θα χρησιμοποιήσει αυτό το χρόνο και τις δυνατότητε που έχει μέχρι τις 31 Μαρτίου που θα κλείσει οριστικά η αντιπροσωπεία της ΟΑΣΕ στην Λευκορωσία και θα προσπαθήσει η Λιθουανία να βρει κάποια πρέπουσα λύση για το πρόβλημα αυτό μέσα στο πλαίσιο αυτό η Λιθουανία ως προεδρεύουσα της ΟΑΣΕ ζητά και από τις ε, όμορες χώρες να υπάρξει συνεργασία και από όλη την, την διεθνή κοινότητα και ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να υπάρξει ε, συνειδητοποίηση της θέσης της διεθνούς κοινότητας στο Μίνσκ για να σταματήσει η πίεση στην κοινωνία των πολιτών, οι παράνομες ε, έρευνες και κρατήσεις και ως ε, προεδρεύουσα χώρα της ΟΑΣΕ η Λιθουανία υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίλυση των προβλημάτων στη Λευκορωσία και ήδη ο πρόεδρος και ο, της κοινοβουλευτικής ε, συνέλευσης ΟΑΣΕ και ο υπουργό μας ζήτησαν να υπάρξει μια συζήτηση με τον κύριο Μαρτίνοφ και του ζήτησαν να απελευθερώσει τους κρατούμενους και τους δημοσιογράφους αμέσα έχει επίσης ε, εκδηλώσει η ΟΑΣΕ την ε, θέλησή της να παρακολουθήσει από κοντά τις δίκες οι οποίες θα λάβουν χώρα στη Λιθου... στην ε, Λευκορωσία στο άμεσο μέλλον. Παροτρύνουμε επίσης τη την Λευκορωσία να έρθει σε επαφή με επικοδομητικό τρόπο με τις αρχές της ΟΑΣΕ και να τηρήσει τις διεθνές, διεθνείς υποχρεώσεις της Λευκορωσίας. Ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η παρουσία της αντιπροσωπείας της ΟΑΣΕ οποίος Θέλουμε λοιπόν να υπάρξει μια έστω ελάχιστη διαθεσιμότητα από την πλευρά της Λευκορωσίας να συνεχίσουν οι ενέργειες της ΟΑΣΕ. Θα ήθελα να σα ζητήσω, κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ζητήσει από τη Λευκορωσία να ε, να ανακαλέσει αυτή την απόφαση για το κλείσιμο του γραφείου της ΟΑΣΕ, γιατί είναι απαραίτητη η παρουσία της ΟΑΣΕ στη Λευκορωσία και είναι απαραίτητο οι αρχές Λευκορωσίας να απελευθερώσουν τους πολιτικούς κρατουμένους και όλους αυτούς οι οποίοι κρατούνται για πολιτικούς λόγους. Τέλος, θα πρέπει να υπάρχει υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών της Λευκορωσίας, θα πρέπει να γίνει πιο ισχυρή και πιο ορατή η χρηματοδότησή μα θα πρέπει να ανακατευθυνθεί για να βοηθήσει την κοινωνία των πολιτών και να εξασφαλίσει καλύτερη επαφή σε επίπεδο απλών ανθρώπων. Θα πρέπει να οργανωθεί και μια διάσκεψη χορηγών τον ε, ε, Φεβρουάριο και το Πανεπιστήμιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βίλνιους θα πρέπει να αντιμετωπίσει και ένα νέο κύμα από φοιτητέ και διδάσκοντες οι οποίοι κινδυνεύουν να εκδιωχθούν από την Λευκορωσία. Χαιρόμαστε λοιπόν για την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και προσδοκούμε σε περαιτέρω ε, ενέργειες από τη δική σας πλευρά για την ενίσχυση του Πανεπιστημίου του Βίλνιους. <clears throat> Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να δείξουμε στην κοινωνία των πολιτών της Λευκορωσίας ότι θα υπάρξει υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό μπορεί να γίνει με διευκόλυνση της, παρα... της παροχής ε, προξενικών θεωρήσεων και μείωση των τελών για κάτι τέτοιο. Έχουμε ήδη τονίσει <clears throat> τη σημασία της αντιμετώπισης του θέματος αυτού ως Λιθουανία προς τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρέπει όποιες, οποιοδήποτε φράγμη να μην θίξουν τους πολίτες της ε, Λευκορωσίας οι οποίοι θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ταξιδέψουν σε χώρες που έχουν κράτος δικαίου και δημοκρατικές ελευθερίες και να νιώσουν σαν ένα πραγματικό κομμάτι της ε, Ευρώπης. Και αξίζει όλη αυτή την υποστήριξη ο λαός Λευκορωσίας. Ευχαριστώ κύριε Υφυπουργέ. Ο κύριος Φίλε, ο Επίτροπος, έχει το λόγο. Uh, κύριε Πρόεδρε, κύριοι Πρόεδροι, αγαπητοί συνάδελφοι, θα σας ευχαριστήσω πρώτα εσάς και του συναδέλφους σας για τις προσπάθειές σας και κυρίως για την διοργάνωση πρόσκληση δηλαδή των ε, σημαντικών αυτών προσωπικότητων και διοργάνωση της ε, ε, παρούσας συνεδρίασης. Η Λευκορώσοι είναι φίλοι μας, γείτονες και εταίροι μας και τις σκέψεις μας θα πρέπει να εμπνέει η ανάγκη προστασίας των συμφερόντων τους με ανοιχτή ανταλλαγή απόψεων για την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε. Ακριβώς αυτό απαιτείται. Ελπίζω η σημερινή συζήτηση να αποτελέσει φάρο για, την, για τον προσανατολισμό των σκέψεών μας για το πώς θα προχωρήσουμε από τούδε και στο εξή. Ο χρόνος δεν είναι με το μέρος μας. Πρέπει να αντιδράσουμε ταχύτατα στα γεγονότα του Δεκεμβρίου και να συζητήσουμε την ενδεχόμενη αντίδρασή μας με τις χώρες μέλη. Ωστόσο, εκφράζω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι είμαστε σε θέση να μοιραστώ μαζί σας και την αξιολόγηση που κάνουμε της καταστάσεως καθώς και τις ε, δράσεις που προτείνουμε να αναλάβουμε ε, βραχυπρόθεσμα. Η άποψή μου είναι ότι έχουμε καθήκον να δράσουμε ταχαίως και με τρόπο ανάλογο. Και αυτό πρέπει να το πράξουμε χωρίς να απομονώσουμε τους λευκορώσους πολίτες. Για τους λόγους αυτούς επιθυμώ να τονίσω την θεμελιώδη ανάγκη μιας ισορροπημένης προσέγγισης που θα σημάνει περισσότερο άνοιγμα απέναντι στους πολίτες και στην κοινωνία των πολιτών με ταυτόχρονα παράλληλα στοχευμένα μέτρα κατά των λευκορωσικών αρχών και με επανεξέταση των κυρώσεων. Χωρίς να αποδυναμώσουμε την ανταπόκρισή μας, την αντίδρασή μας, αλλά με ε, συγκεκριμένη στόχευση για βελτίωση μάλλον παρά ε, δυσχέρανση της ζωής των πολιτών. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε ανοιχτούς τους διάβλους άμεσης χορήγησης βοήθειας σε μη κρατικέ οργανώσεις, στα μέσα ενημέρωσης και στους ε, φοιτητέ. Μέτρα για την βελτίωση της κινητικότητας των λευκορώσων πολιτών που επιθυμούν να μεταβούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρώ ότι συμφωνούμε όλοι στην αξιολόγηση της σημερινής κατάστασης. Ήταν βαθύ το σοκ που υπέστημεν μετά από τα γεγονότα της 20ης Δεκεμβρίου. Συμφωνούμε με την άποψη του ΟΑΣΕ ότι η Λευκορωσία δηλαδή έχει ακόμα πολύ δρόμο να κάνει για να ανταποκριθεί στις υποχρώσεις που της επιβάλλει η συμμετοχή της στον ΟΑΣΕ. Επίσης η εκλογική διαδικασία αμαυρώθηκε από τις κρατήσεις που επευλήθηκαν σε βάρος εκπροσώπων της αντιπολίτευσης. Περίπου 700 άτομα κρατήθηκαν τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Οι περισσότεροι απολύθηκαν από τα κρατητήρια. Ορισμένοι και μάλιστα υποψήφοι στις προεδρικές εκλογές αντιμετωπίζουν τώρα κατηγορίες που ενδέχεται να τους οδηγήσουν για 15 χρόνια στη φυλακή η Κάθριν Άστον, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είπατε εκπρόσωπος, καταδίκασε τις ενέργειες αυτές και ζήτησε από τις ε, λευκορωσικές αρχές να απολύσουν όλους όσοι κρατούνται για τους λόγους αυτούς. Σε κοινή δήλωση με την Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Χίλαρη Κλίντον. Η κράτηση ειρηνικών διαδηλωτών εξακολουθεί να είναι απαράδεκτη και η απόλυσή τους είναι η νούμερο ένα προτεραιότητά μας. Έχοντας τώρα εξηγήσει την θέση μας, θεωρώ ότι το επόμενο βήμα θα πρέπει να είναι να καθοριστούν ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν απέναντι στη Λευκορωσία. Η λήψη της απόφασης αυτής, όπως είπα και προηγουμένως, θα πρέπει να βασίζεται σε μια εξέβρεση ισορροπίας ανάμεσα σε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τις λευκορωσικές αρχές σχετικά με τον αποτροπιασμό μας και την καταδίκη των ε, ενεργειών τους και από άλλη ένα μήνυμα υποστήριξης προς το λευκο, λευκορωσικό λαό. Αυτό θα πρέπει να μην οδηγήσει σε απομόνωση του λευκορωσικού λαού όπως είχε γίνει με μέτρα που λύθηκαν πριν από το 2008 θα πρέπει να διακριθούν τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν κατά προτεραιότητα από άλλα τα οποία θα χρειαστούν περαιτέρω ε, σχεδιασμό. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι μια προσέγγιση σε δύο φάσεις. Πρώτα θα ήθελα να σας ενημερώσω κύριε Πρόεδρε και τους άλλους παρόντες εδώ για την πρώτη φάση της αντιδράσεώς μας, δηλαδή τα μέτρα προτεραιότητας. Η εισαγωγή ε, απαγόρευσης έλευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε βάρος του πρόεδρου Λουκασένκο και άλλων μελών της κυβέρνησης του αυτό είναι μια πρώτη επιλογή. Άλλες επιλογές θα συζητηθούν στο, στη συνέχεια μάλλον των αποφάσεων του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της 1ης Ιανουαρίου. Πρέπει να εξετάσουμε τον καλύτερο τρόπο επιβολής κυρώσεων ώστε να είναι εξασφαλισμένο το αποτέλεσμά τους. Ο στόχο μα είναι βεβαίω να επιτύχουμε την απόλυση των πολιτικών κρατουμένων, καθώς και την ασφάλεια όλων όσοι εξακολουθούν να κρατούνται. Το μήνυμά μας προς το Μίνσκ είναι ξεκάθαρο. Η Λευκορωσία θα πρέπει αμέσως να απολύσει τους κρατουμένου και να πάυσει την ποινική δίωξη των δημοκρατικών δυνάμεων, εάν επιθυμεί να αποφύγει τις κυρώσεις. Το χρονοδιάγραμμα των απολύσεων αυτών θα πρέπει να είναι της τάξης ωρών ή ημερών, όχι εβδομάδων. Πέρασα το μήνυμα αυτό στον Υπουργό Εξωτερικών Μαρτίνοφ και η κάθε Άστον επέμεινε στην, ε, ε, στο επίγον της κατάστασης στη συνάντησή της μαζί του. Θα έρθω τώρα στα θετικά μέτρα και κυρίως εκείνα τα οποία θα απευθύνονται στην κοινωνία των πολιτών. Η η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσεω σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συντάξει επιλογές επιγόντων μέτρων με στόχο μη κρατικέ οργανώσεις, μέσα ενημέρωσης και φοιτητέ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βεβαίω έχει και αυτό την δυνατότητα να προσφέρει υποτροφίες σε σπουδαστές οι οποίοι εκδιώχθηκαν από τα πανεπιστήμια. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συνενώσουμε τις προσπαθίες μας εν προκειμένου. Τονίζω ότι ενθαρρύναμε και τις χώρες μέλη να κάνουν παρόμοια εγχείρημα, να προβούν σε παρόμοιο εγχείρημα επανεξέτασης. Επίσης, η συνάντηση στις 2 Φεβρουαρίου της ομάδας των δωρητών υποστηρίζει την ε, πρόταση αυτών των χωρών μελών η διευκόλυνση χορήγηση προξενικών θεωρήσεων επίσης πρέπει να παραμείνει ε, ως προτεραιότητά μας. Βεβαίως θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτό δεν θα αποτελέσει δώρο προς, τους, προς τις αρχές. Θα χρειαστεί συντονισμένη δράση των ε, προξενείων των χωρών μελών στο Μίνσκ. Κυρίε και κύριοι, στρέφοντας τα βλέμματα στο μέλλον, στην δεύτερη φάση δηλαδή της ε, ανταπόκρισης μας στα γεγονότα αυτά, θα ήθελα να μοιραστώ ορισμένες σκέψεις μου για ορισμένες άλλες πτυχές του θέματος. Σχετικά με το κοινό ενδιάμεσο πρόγραμμα, νομίζω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε, χωρίς να καταλήψουμε το σχέδιο ωστόσο, αλλά να διαβολευτούμε με την κοινωνία των πολιτών, και αν είναι απαραίτητο να επανεξετάσουμε το περιεχόμενο του Joint Interim Plan. Είναι πιο σημαντικό ακόμη σήμερα από το παρελθόν οι πολίτες της Λευκορωσίας να έχουν πλήρη εικόνα των προσφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε ό,τι αφορά την υποστήριξη της ΕΝΠΗ στη Λευκορωσία, δηλαδή της πολιτικής γειτονίας αυτό θα σημάνει διοχέτευση βοήθειας συγκεκριμένα στοχευμένης στην κοινωνία των πολιτών. Εν τέλει, κύριε Πρόεδρε και εσείς αγαπητοί συνάδελφοι, πιστεύω ότι η Λευκορωσία πρέπει να συνεχίσει να συμμετέχει στην ε, πολιτική ανατολικής γειτονίας. Η συμμετοχή της μέχρι τώρα ήταν περιορισμένη και δεν συνεπάγεται σημαντική οικονομική ε, ενίσχυση αλλά είναι σημαντικό η παρούσα κρίση να γίνει αντικείμενο διαχείρισης στο σωστό περιφερειακό πλαίσιο και το βάρος άλλων σημαντικών εταίρων να χρησιμοποιηθεί πλήρως Αυτά σημαίνουν βέβαια δύσκολο εγχείρημα ισορροπίας. Θα πρέπει να παρακολουθούμε την εξέλιξη των γεγονότων διαρκώς. Ελπίζω ότι μπορώ να υπολογίζω στην υποστήριξη των Ευρωβουλευτών και των άλλων ενδιαφερομένων μερών και αναμένω με ενδιαφέρον την έκφραση των δικών σας απόψεων. Ευχαριστώ. Eh, Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Θα δώσω τώρα το λόγο στους ε, τρεις ε, προέδρους ε, που με συνοδεύουν σε αυτήν τη συνεδρίαση. Πρώτα θα δώσω το λόγο στην κυρία Χαούταλα, πρόεδρο της Υποπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θέλω να αποτίσω φόρο τιμή στην κοινωνία των πολιτών στη Λευκορωσία και τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί ήδη για να μπορέσει να δοθεί μια σωστή πληροφόρηση και υλικό για μια ενδελεχέστερη έρευνα σε σχέση με τα γεγονότα της 19ης Δεκεμβρίου και στη συνέχεια. Όπως τόνισαν πολλοί ομιλητέ από την Λευκορωσία και από την Κομισιόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μια πιο ενεργή και πιο στενή σχέση με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην Λευκορωσία και με τη δημοκρατική αντιπολίτευση στη χώρα αυτή και πρέπει να αναγνωρίσουμε την ανάγκη να γνωρίσουμε ποια είναι η πραγματικότητα σε σχέση με τους αλληλοσυγκριόμενους συγκρόμενους ισχυρισμούς για το ποιος ήταν υπεύθυνο για τις βίες ενέργειες της 19 9η Δεκεμβρίου που είναι φυσικά και η βάση για τι καταγγελίε και τι κατηγορίε εναντίον εκατοντάδων ειρηνικών διαδηλωτών στη χώρα αυτή. Θέλω επίση να εξασφαλίσω ότι η κοινή δήλωσή μα μετά από τη σημερινή συζήτηση θα συμπεριλαμβάνει και την έκκληση του Υπουργού Εξωτερικών Σεβίτσιους ότι θα ζητήσουμε από τις αρχές Λευκορωσίας να ε, ακυρώσουν την απόφασή τους να κλείσουν τα γραφεία της ΟΑΣΕ γιατί, στην Λευκορωσία στο Μίνσκ. Γιατί πιστεύω ότι η ΟΑΣΕ μαζί με τις ε, υπηρεσίες του ΟΗΕ μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο παρακολούθησης της κατάστασης εκεί και επίσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να πράξει το ίδιο με μια δική του αποστολή. Ευχαριστώ κύριε Άουταλα. Ο κύριος Προτεσίεβιτς έχει το λόγο, πρόεδρος αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τη Λευκορωσία. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θέλω καταρχήν να κάνω μια αναφορά σε αυτά που είπε ο πρεσβευτής κύριος Άρενς στην ε, αρχική του παρέμβαση ότι οι πρόσφατες εκλογές της Λευκορωσίας δεν είναι οι πρώτες τέτοιες εκλογές όπου παρατηρήθηκε έλλειψη αμεροληψίας και έλλειψη σωστής διαδικασίας καταμέτρησης των ψήφων που φυσικά είναι μια κεντρική προ... πρώτερη απέτηση για οποιασδήποτε δημοκρατικές εκλογές. Η αντιπροσωπεία τη οποία έχω την τιμή να προείσταμε είναι η μόνη αντιπροσωπεία μεταξύ των αντιπροσωπείων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δεν έχει διακοινοβουλευτική διάσταση. Διότι λόγω της συνεχιζόμενης αντιδημοκρατικής διακυβέρνησης στη Λευκορωσία εμείς εστιάζουμε την προσοχή μας στην επαφή και τη συνεργασία με τη δημοκρατική αντιπολίτευση και την κοινωνία των πολιτών. Δεν έχουμε όμως αντιταχθεί στη νέα πρόταση της Κομισιόν και του Συμβουλίου να αναπτύξουμε μία μορφή διαλόγου με την κυβέρνηση της Λευκορωσίας για να μπορέσουμε να επιτύχουμε ουσιαστικές αλλαγές και σε οικονομικό και σε δημοκρατικό επίπεδο στη Λευκορωσία. Μετά όμως τα γεγονότα της 19ης και 20ης Δεκεμβρίου πέρσι, είναι πεποίθησή μου και ελπίζω ότι και τα μέλη της αντιπροσωπείας μου συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις με μένα, πιστεύω ότι δεν υπάρχει περιθώριο για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση Λευκορωσίας σαν να μην συμβαίνει τίποτα, σαν να είναι μια φυσιολογική πορεία πραγμάτων. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε και άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον τον Επίτροπο κύριο Φίλε, αυτό το οποίο χρειαζόμαστε <clears throat> είναι να απαιτήσουμε την απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων και των υπολείπων συλληφθέντων και επίσης να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξουν πραγματικά αποτελεσματικά μέτρα για να αρρωγήσουν τη δημοκρατική αντιπολίτευση και την κοινωνία των πολιτών στη Λευκορωσία, τι μη κυβερνητικέ οργανώσει, του ακτιβιστέ, τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωση, για να ενισχυθεί η κοινωνία των πολιτών στη Λευκορωσία. αυτό είναι και ο μόνο τρόπο με τον οποίο μπορεί η χώρα αυτή να γίνει πιο δημοκρατική. Και η δημοκρατία καθώ και η ελευθερία είναι οι αξίε τις οποίες ενστερνίζονται και θέλουν να πραγματοποιήσουν και οι πολίτες της Λευκορωσίας. Η Λευκορωσία είναι ένας <clears throat> εγκύτατος γείτονα μας <clears throat> και θα πρέπει να βρούμε ένα νέο τρόπο να πλησιάσουμε τους πολίτες αυτής της χώρας. Ο κύριος Βιγγένιν, πρόεδρος της Euronest. Δύο λεπτά κι εσείς σας παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι. Η Ανατολική Γειτονία ξεκίνησε για να βελτιώσει τη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των έξι χωρών και αυτή στιγμή ξεκίνησε πέντε από τις χώρες αυτές με διάφορα πάνω και κάτω μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν τους νέους μηχανισμούς για να ε, εργαστούν επί των κυριότερων τομέων αυτής της ε, ε, συνεργασίας με κυρίως βελτίωση της δημοκρατίας, σεβασμού ανθρώπινων δικαιωμάτων κλπ. και κράτους δικαίου. Μία από τις χώρες αυτές δεν μπόρεσε να δείξει επαρκή δέσμευση στους στόχους που μόλις ανέφερα και για αυτό το λόγο δεν μπορέσαμε να αρχίσουμε πραγματικό κοινοβουλευτικό διάλογο και συνεργασία με τις λευκορωσικές ε, αρχές είτε διμερή είτε πολυμερή, σε πολυμερές πλαίσιο δηλαδή. Ελπίζουμε οι ε, εκλογικές, ε, οι προεδρικές εκλογές του χρόνου αυτού να ελπίζαμε μάλλον οι προεδρικές εκλογές που έγιναν θα μας επέτρεπαν να κάνουμε μια νέα φετηρία και η προεκλογική εκστρατεία μας έδινε κάποιο θάρρος προς την κατεύθυνση αυτή, έστω και αν θεωρούσαμε ότι οι βελτιώση που είχαν γίνει ήταν μάλλον καλοπιστικού χαρακτήρα, αλλά βλέπαμε κάποια κίνηση. Ωστόσο, δυστυχώς η 19η και 20η Δεκεμβρίου κατέστρεψαν τις ελπίδες αυτές και ε, μας προκάλεσαν σημαντικές αμφιβολίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα της πολιτικής μας απέναντι στη Λευκορωσία. Το ερώτημα που τίθεται τώρα είναι τι θα πρέπει να αλλάξει. Δεν θα πρέπει να βιαστούμε πολύ στις αποφάσεις μας, γιατί οι βιαστικές αποφάσεις δεν είναι απαραίτητα καλές αποφάσεις. Νομίζω ότι θα πρέπει να αποφύγουμε να τιμωρήσουμε των εισαγωγικών το λευκορωσικό λαό για πράγματα για τα οποία ευθύνονται ο πρόεδρος και οι αρχές. Χρειαζόμαστε πιο καλά στοχευμένε κυρώσει, αλλά και πιο καλά στοχευμένη υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών και των ανθρώπων εκείνων που προσπαθούν να επιτύχουν εκδημοκρατισμό της ε, λευκορωσικής κοινωνίας. Αυτά θα τα συζητήσουμε και στην επόμενη, ε, την επόμενη εβδομάδα, στην περίοδο συνόδου του Στρασβούργου και ελπίζω θα μπορέσουμε να προτείνουμε καλές λύσεις στο Συμβούλιο των Υπουργών. Χωρίς να πέσουμε σε ιστέρια, πρέπει ωστόσο να είμαστε πολύ ξεκάθαροι και επίμονοι σε δύο βασικά θέματα απόλυση όλων των κρατουμένων από τη 19η και 20η Δεκεμβρίου και άρση της δίωξης των προσώπων που συμμετείχαν σε διαδηλώσεις. Άλλα θέματα όπως η αποδοχή ε, της, της μετάβασης μιας διεθνούς επιτροπής η οποία θα εξετάσει τα ε, γεγονότα θα πρέπει να ε, γίνει με πίεση προς τον Πρόεδρο και τις αρχές. Τέλος, θα πρέπει όλα τα θεσμικά όργανα να τηρήσουν μια κοινή γραμμή ώστε να επιτύχουμε τον απότερο στόχο μας, δηλαδή μια δημοκρατική Λευκορωσία. Εάν δεν υπάρξει κοινή γραμμή δεν θα επιτύχουμε και ε, θα, ε, αποτελέσματα. Αρχίζει τώρα η πραγματική συζήτηση με την ε, τοποθέτηση πρώτα των συντονιστών που και αυτοί θα πρέπει να μιλήσουν πέντε λεπτά ούτως ώστε όλοι να μπορέσουν να μιλήσουν στη συνέχεια. όπως επίσης ε, και οι ομιλητές μας να μπορέσουν να απαντήσουν. Σας παρακαλώ να αναφερθείτε και στις συστάσεις που θα πρέπει να δώσετε για τις δράσεις της Ένωσης και πιο συγκεκριμένα την εντολή για την αποστολή ad hoc στην ε, Λευκορωσία. Ο κύριος Μπρόκ, συντονιστής του ΕΛΚ, δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, εξ ονόματος της ε, Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Λαϊκού Κόμματος ευχαριστώ για άλλη μια φορά τους εκπροσώπους της Λευκορωσίας καθώς και τους υπολείπους εκπροσώπους της Κομισιόν καθώς και των υπουργοεξωτερικών της Λιθουανίας για την ενημέρωση που μας έκαναν. Σήμερα έλαβα επιστολή του Λευκορώσου πρέσβη στο Βερολίνο. Μου γράφει ότι εάν ψηφίσουμε επικριτικό ψήφισμα κατά τη Λευκορωσία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τότε πλέον η Λευκορωσία δεν θα έχει άλλη δυνατότητα παρά να συνεργαστεί στενότερα με τη Ρωσία. Αυτά μου φαίνονται εμένα απειλές απαράδεκτες. Γιατί τα θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων, δημοκρατίας και κράτους δικαίου δεν είναι διαπραγματευτά. Για το λόγο αυτό πρέπει να δούμε πώς θα δράσουμε, πώς θα εκφραστούμε κριτικά, πώς δεν θα δεχθούμε τα όσα συνέβησαν και ποιους μηχανισμούς θα υιοθετήσουμε. Αν θα πάει τώρα μια ειδική αντιπροσωπεία εκεί, αυτό θα προτιμήσω να μου το πούν οι Λευκορώσοι φίλοι μας. Εάν θεωρούν ότι κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει, τότε εγώ θα είμαι υπέρ. Αλλά νομίζω αυτό πρέπει να το κρίνουν οι ίδιοι και να εμείς να ακολουθήσουμε τη συμβουλή τους δεν θεωρώ ότι μπορώ εγώ να λάβω την τελική απόφαση. Το δεύτερο είναι τα μέτρα. Χάρηκα για τα όσα άκουσα από τον Επίτροπο Φούλε. Είπε μεταξύ άλλων ότι οι αποφάσεις που θα πρέπει να ληφθούν δεν μπορούν να είναι θέμα μηνών, αλλά μόνο ωρών ή το πολύ ημερών. Και θα είναι καλό, κύριε Επίτροπε, αυτό να μπορέσει να συμφωνηθεί, να μπορέσει να συμμορφωθεί μάλλον με το δικό μας χρονοδιάγραμμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της επόμενης εβδομάδας, όπου μπορούμε τότε ε, να προχωρήσουμε σε μια ακόμα καλύτερη διατύπωση του ψηφίσματός μας. Ψηφίσματός μας. Θεωρώ ότι στα πλαίσια της πολιτικής γειτονίας οι μηχανισμοί και τα μέσα που θα έχουμε στη διαθεσή μας θα πρέπει να είναι τέτοια που να επιτρέπουν περισσότερη δημοκρατική εξέλιξη. Και θα παρακαλέσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεξετάσει το αρχικό σχέδιο που είχαμε τότε περιλάβει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά μας να δίνεται υποστήριξη δηλαδή στην κοινωνία των πολιτών χωρίς να δίνεται υποστήριξη στις αρχές. Τελευταίο, αν όλα αυτά δεν οδηγήσουν σε κάποια πρόοδο θα πρέπει να ξαναδούμε εάν ίσως πρέπει να αναστείλουμε τη συμμετοχή της ε, Λευκορωσίας στην πολιτική ανατολικής γειτονίας. Όχι να την, να την διώξουμε, αλλά να την αναστείλουμε. Διότι, εν πάση περιπτώσει, οφείλει να υποστεί κάποιες συνέπειες η λευκορωσική κυβέρνηση. μεταξύ των ε, αξιώσεων μας θα πρέπει να είναι και η διατήρηση της αντιπροσωπείας, του γραφείου της αντιπροσωπείας του ΟΑΣΕ στο Μίνσκ. Αυτά είναι ολίγη, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μπρόκ. Ο κύριος Σεβερίν έχει το λόγο, συντονιστής των σοσιαλιστών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω καταρχήν να καλωσορίσω όλους τους καλεσμένους μας από τη Λευκορωσία με μεγάλη συγκίνηση. Θα τους χαιρετήσω και εκφράζω την αλληλεγγύη μου μαζί του. Για μένα όλα αυτά είναι κάτι που το έχω ξαναδεί, ένα έργο που το έχουμε ξαναπέξει. Τίποτα καινούριο δεν είναι σε αυτές τις εξελίξεις. Έχουμε την ίδια διάγνωση μαζί σας. Καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να μιλήσουμε με ενιαία φωνή ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμμεριζόμαστε την άποψη ότι το πιο κατεπήγον αυτή τη στιγμή είναι να ζητήσουμε και να επιτύχουμε την απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων. Έλκεται από την κοινή γνώμη ότι προ το παρόν τουλάχιστον δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε το σενάριο του business as usual. Συμφωνούμε επίση ότι και η απομόνωση δεν είναι επιλογή <clears throat> της Λευκορωσίας. Για όλου αυτού του λόγου πιστεύω ότι εφόσον συμφωνούμε με όλα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να προσθέσουμε και την ιδέα ότι στι δικέ μα προσπάθειε θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι και με τους άλλους εταίρους της Λευκορωσίας, τις γειτονικές της χώρες που είναι εταίροι και σύμμαχοί μας και με τους οποίους είμαστε στα πλαίσια διαπραγματεύσεων διαφόρων συμφωνιών και ομιλώ για την Ουκρανία και τη Ρωσία, θα πρέπει να ακολουθηθεί μια κοινή γραμμή από όλους. Κατά τα άλλα, τι μπορούμε να πούμε, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι όλα έχουν ελεγχθεί. Πρέπει να κινητοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις μας για να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας θα πρέπει να κατανοήσουμε τι δεν μπορούμε να κάνουμε και πρέπει να έχουμε και την υπομονή και την σοφία να καταλάβουμε τι είναι πρόσφορο να γίνει και τι δεν είναι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σεβερίν γιατί σεβαστήκατε το χρόνο ομιλίας. Η κυρία Ογιολάντα για δύο λεπτά εξ ονόματος φιλελεύθερης και δημοκρατικής ομάδας θέλω να εκφράσω και εγώ την ειλικρινή μας ε, υποστήριξη και τις ευχές μας προς το λαό της Λευκορωσίας την συμπαράστασή μας σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση. Είμαστε εδώ για να επανεξετάσουμε τη σχέση μας με το τωρινό καθεστώς της Λευκορωσία. Όσο λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε μία ενιαία στάση, το μήνυμά μας ήταν πάντα ακουστό. Τώρα όμως πρέπει να περάσουμε και στο διατάφτα και όχι απλώς να παραμείνουμε σε επίπεδο φραστικών ε, δηλώσεων. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να έχουμε την ε, εταιρική σχέση μέσα στα πλαίσια της ε, ανατολικής πολιτικής γειτονίας με τη Λευκορωσία όσο υπάρχουν κρατούμε στις φυλακές. Έχουμε δει ότι οι πολιτικές του μαστιγίου και του καρότου, όπως λένε οι Αγγλοσάξονες, ότι δεν έχουν λειτουργήσει. Έχουμε ακόμα το ίδιο καθεστώς και ένα καθεστώς το οποίο είναι απάνθρωπο και αυταρχικό. Πρέπει να τονίσουμε σαφώς ότι πρέπει να υπάρξει αλλαγή καθεστώτος. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος προς τον οποίο θα εργαστούμε όλοι από κοινού και μαζί με την αντιπολίτευση της Λευκορωσίας και μαζί και με το λαό της Λευκορωσίας. Το κυριότερο όπλο μας στην εξωτερική πολιτική το ξέρουμε σαν πολιτική είναι πάντα οι κυρώσει. Και η ομάδα η φιλελεύθερη υποστηρίζει μια σειρά κυρώσεων που ξεκινούν από την άρση προξενικών θεωρήσεων και από το πάγωμα οικονομικών διευκολύσεων προς τη χώρα αυτή, λαμβάνοντας όμως πάντα στα πλαίσια αυτά τις ανάγκες των απλών <clears throat> πολιτών των μέσων ενημέρωση, την ανάγκη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, επίση τη ανάγκη να υπάρξει μια μεγαλύτερη φιλελευθερωποίηση των δυνατοτήτων ταξιδίου για του απλού πολίτε και φυσικά για την υποστήριξη των φοιτητών οι οποίοι επλήγησαν λόγω τη πολιτική του δραστηριότητας στα Πανεπιστήμια τη Λευκορωσίας. Τέλο, και όχι τελευταίο, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν θα πρέπει να παραγνωρίσουμε και το ρόλο της Ρωσίας στην τωρινή κατάσταση στη Λευκορωσία ιδίω μετά από τις ε, δηλώσεις που ακούσαμε αμέσως μετά από τις εκλογές του Δεκεμβρίου από τον πρόεδρο Μετβέντεφ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σούλτς, εξ ονόματος των Πρασίνων, για δύο λεπτά. Αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητοί φίλοι από τη Λευκορωσία, επανέρχομαι σε αυτό που είπε ο πρόεδρός μας, κύριος Μπούσεκ, ότι βρισκόμαστε σε ανοιχτή διαβούλευση σχετικά με το τι θα κάνουμε μετά από αυτή την ε, βάρβαρη νοθεία των εκλογικών αποτελεσμάτων. Και ε, νομίζω ότι οι πιο σημαντικές αξιώσεις ξεκαθαρίστηκαν, δηλαδή απόλυση των κρατουμένων, μάλιστα και αποζημίωσή τους, απόσυρση των παράλογων κατηγοριών, θα πρέπει να ιδρυθεί και εξεταστική επιτροπή για την ίδια την εκλογική νοθεία, θα χρειαστεί δεύτερος γύρος εκλογών, διότι προφανώς δεν επετεύθη από πλευρά Κασένκο το 50% των ψήφων, θα πρέπει να ανοίξει πάλι το γραφείο του ΟΑΣΕ, να διευκολυνθούν οι προξενικές θεωρήσεις. Νομίζω σε αυτόν τον κατάλογο μέτρων είμαστε όλοι σύμφωνοι. Γι' αυτό θα έρθω λίγο περισσότερο τώρα στους στρατηγικούς στόχους, γιατί από την δική μου εμπειρία στην αντικομουνιστική αντίσταση στην ε, προανατολική Γερμανία. Γνωρίζω πώς αντιμετωπίζουν, πώς αντιδρούν οι δικτάτορες όταν στριμωχτούν στη γωνία. Κάνουν ακόμα πιο βάρβαρα καταπιεστικό το σύστημά τους. Γι' αυτό εγώ θα έλεγα να δώσουμε ειδική εντολή στην Λέβη Άστον να πάει στο Μίνσκ να θέσει ξεκάθαρα τις αξιώσεις και απαιτήσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ανακοινώσει τις ε, κυρώσεις που θα επιβληθούν στον Λουκασένκο εάν δεν συμμορφωθεί. Σε ό,τι αφορά τώρα την απαγόρευση έλευση εδώ του Λουκασέρκο, τέτοια πράγματα τα είχαμε και πριν. Δεν τον απασχολούν τόσο πολύ. Εάν δεν περιλάβουμε στα μέτρα αυτά ολόκληρο το καθεστώς Λουκασένκο. Να μην επαναλάβουμε τα λάθη που κάναμε παλαιότερα με τη Ρωσία όταν έπρεπε να είχαμε αντιδράσει απέναντι στον Πούτιν. να χρησιμοποιήσουμε την ειδική διάσκεψη ε, που θα γίνει την άνοιξη στη Βουδαπέστη για την Ανατολική Γειτονία για να προσκαλέσουμε τον Λουκασένκο μέχρι τότε λοιπόν να μην του επιβληθεί απαγόρευση προξενικής θεώρησης για να του θέσουμε τα θέματα, να τον αναγκάσουμε να μιλήσει και να δείξει το πραγματικό του πρόσωπο. Ευχαριστώ κύριε Σούλτς, ο κύριος ε, Τάνοκ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, εξ ονόματος της ομάδας των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών και εγώ θέλω να σας χαιρετήσω σε αυτή τη συζήτηση και να σας καλωσορίσω. Εγώ δεν εκπλήσωμαι από αυτά τα οποία γίνονται. Μετράνε περισσότερο τις διμερεί σχέσεις οι Λευκορώσοι και όχι τι σχέσει του με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη φορά τα πράγματα όμω πρέπει να είναι διαφορετικά. Αυτή τη φορά θα πρέπει η ΟΑΣΕ να ε, λέγανε θα έπρεπε η ΟΑΣΕ αυτή τη φορά να επικυρώσει τα αποτελέσματα των εκλογών. Αλλά δεν μπορούν να προβλέψουν ούτε και οι αξιωματούχοι της ε, Λευκορωσίας την παράδοξη πολλές φορές και αλλοπρόσαλη συμπεριφορά του Λουκασέγκο, ο οποίος παραμένει ο όμος Σοβιέτικος της περιοχής. Προσπαθούν με λαθροχειρίες να επιτύχουν μία ανοθεία για το εκλογικό αποτέλεσμα και αν αυτό δεν γίνεται χρησιμοποιούν βία μέτρα κατά των εκπροσώπων της αντιπολίτευσης. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να ζητήσουμε από την ύπατη εκπρόσωπο να επιμείνει στεναρά στο να υπάρξει απελευθέρωση όλων των δημοκρατικών αγωνιστών και κρατουμένων και η επανάληψη των προεδρικών εκλογών. Συμφωνώ απόλυτα με τους πράσους. Τα ίδια έγιναν και στην περίπτωση των ε, Ουκρανικών εκλογών της Πορτοκαλή Επανάσταση, και εάν είναι πραγματικό συνταγματικό δικαστήριο, συνταγματικό δικαστήριο της Λευκορωσίας θα πρέπει να επιμείνει στην επανάληψη των εκλογών. Και αυτή η επανάληψη θα πρέπει να τηρεί όλες τις προϋποθέσεις της, ΟΑΣΕ και έχουμε φυσικά μια μεγάλη αποστολή για την παρακολούθηση των εκλογών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα και αν τα απορρίψει αυτά όπως είναι πολύ πιθανό το Μίνσκ θα πρέπει να προχωρήσουμε σε ευφυείς κρατήσει, ε, κυρώσεις όχι εναντίον του λαού αλλά εναντίον των ηγετών με παγώματα στοιχείων των ενεργητικού του κτλ. Και φυσικά το κόμμα μου υποστηρίζει και μια αντιπροσωπεία ad hoc εάν θεωρεί η δημοκρατική αντιπολίτευση στην Λευκορωσία ότι θα είναι πρόσφορη. Πρέπει όμως να ρωτήσω πόσο καιρό ακόμα μπορούμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δεχόμαστε μια κουβανικού χαρακτήρα δικτατορία στην καρδιά της Ευρώπης. Ευχαριστώ κύριε Τάνοκ, ο κύριος Σόλτσε, εξ ονόματος της για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί φίλοι από τη Λευκορωσία, αρχές Δεκεμβρίου στο Παρίσι διεξήχθη συνέδριο της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και έχουμε και την διακήρυξη εδώ της Δημοκρατικής Αντιπολίτευσης της Λευκορωσίας. Ο Σεργέη Καριάκιν τότε στη διάσκεψη αυτή που είπα προηγουμένως είχε φανεί αισιόδοξο ότι θα μπορούσε να προχωρήσει ένας εκδημοκρατισμός. Γνωρίζουμε βέβαια από την έκθεση της ΟΑΣΕ πώς πήγαν τα πράγματα. Η δική μας πολιτική ομάδα, η Ενωτική Αριστερά, είναι απολύτως της γνώμης ότι θα πρέπει να υιοθετηθούν οι αξιώσεις που ζήτησαν και οι υπόλοιποι εδώ, δηλαδή απόλυση των κρατουμένων, ε, όχι κλείσιμο του γραφείου του ΟΑΣΕ. Πάλι τον Νοέμβριο είχαμε ψηφίσει ψήφισμα για την παραπέρα δράση του ΟΑΣΕ και αυτό θα πρέπει να τηρηθεί. Θα επανέλθω στα λόγια του κ. Μιλίνκεβιτς που είπε ότι από τη Σκοπιά της ε, λευκορωσικής αντιπολίτευσης είναι απαραίτητο να επανεξεταστεί η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αρχές αυτές που πιστεύουμε όλοι είναι η ανοχή και μεταξύ άλλων και η ε, αξιοπιστία της πολιτικής. Αμφιβάλλω και εδώ συμφωνώ με τον προαναλύσαντα Σούλτς ότι θα πρέπει να βάλουμε τώρα ένα σύρτη στην περαιτέρω πορεία της Λευκορωσίας. Όχι, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τις απόψεις μας απέναντι στον Λουκασένκο, ότι αναμένουμε δηλαδή από αυτόν διόρθωση της πολιτικής του και μετά μπορούμε να συζητήσουμε. Αλλά πρέπει βέβαια να λάβουμε υπόψη κιόλα ότι πολλοί πολίτες και ιδίως στην Λευκορωσική Ήπεθρο ψήφισαν όπως ψήφισαν. Και αυτό πρέπει να μας κάνει να σκεφτούμε ποιες είναι οι ευρωπαϊκές αξίες και πώς περνούν από μας στην ίδια τη Λευκορωσία. Και αυτό θα πρέπει να είναι και μελλοντική αξίωση για την δική μας πολιτική. Δηλαδή η ε, υπεράσπιση των ανθρώπινων και πολιτικών δικαιωμάτων. Ευχαριστώ κύριε Σόλτς. Ο κύριος Μπέλντερ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θέλω. Θα ήθελα κι εγώ να πω ότι είμαι ήδη ότι με απασχολεί ιδιαίτερα η τύχη των πολιτικών κρατουμένων. Εμείς στον Ολλανδικό τύπο διαβάσαμε άρθρα, ε, τρομακτικά άρθρα για, την, ε, για το μέγεθος της καταστολής ε, στην Λευκορωσία. Αυτή η δική μας αντίδραση θα βοηθήσει πραγματικά τους Λευκορώσους. Εγώ την προηγούμενη εβδομάδα είχα επαφές με κόσμο από το Μίνσκ και η κοινωνία των πολιτών είναι ιδιαίτερα συντετριμένη από αυτά τα γεγονότα. Αλλά όμως και οι πιο φιλελεύθεροι της κυβέρνησης ε, Λουκασένκο, έχουν ε, σοκαριστεί από όλη αυτή την ιστορία. Πώς θα τους βοηθήσουμε λοιπόν εμείς όλους αυτούς οι οποίοι ανήκουν στον κρατικό μηχανισμό μεν αλλά έχουν ένα πιο ανοιχτό πνεύμα. Δεύτερο, δεν μπορούμε εμείς να απομονώσουμε τη Λευκορωσία και τους ε, πολίτες της δεν θα μπορούσαμε ίσως να αναλάβουμε πρωτοβουλίες για την διαμόρφωση μιας ε, νέας συνείδησης στην κοινωνία των πολιτών, ας πούμε, να μπορέσουμε ε, να έρθουμε σε επαφή με τον κόσμο της υπαίθρου, να έχουμε επαφή με διανομένους, ε, με διάφορα κοινωνικά στρώματα, ούτως ώστε η Ευρώπη να μπορέσει να αντιδράσει ισορροπημένα γύρω από όλα αυτά. Ο κύριος Παλέτσκης είναι ο εισηγητής της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων για την Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Λευκορωσίας η οποία βρίσκεται στο ψυγείο προς την περίοδο, αυτήν την περίοδο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι υπήρξε γενικά μια συνένεση για τις προτάσεις της ε, αντιπολίτευσης στη Λευκορωσία για το πώς να αντιμετωπίσουμε το, τους τα γεγονότα της 19ης και 20ης Δεκεμβρίου και επίσης γύρω από τις απόψεις του κυρίου Φίλε και του κυρίου Γνατάβεβιτς από την Προεδρία της ΟΑΣΕ. Κάποιες κυρώσεις βέβαια είναι αναπόφευκτες μετά τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα. Αυτές οι κυρώσεις όμως θα πρέπει να είναι στοχευμένες και προσεκτικές και θα πρέπει να έχουν σαν στόχο να φέρουν την χώρα και το λαό της κοντύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φυσικά όχι το τρέχον καθεστώς. Όπως είπε ο τουλάχιστον 50% των Λευκορώσων υποστηρίζουν την ευρωπαϊκή κατεύθυνση της χώρας τους. Αν εμεί διαμορφώσουμε σωστά λοιπόν και με ευαισθησία την πολιτική μα έναντι τη Λευκορωσία, μέσα σε ένα-δύο χρόνια μπορούμε να εξασφαλίσουμε να υπάρχει μια ευρεία πλειοψηφία υπέρ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό θα είναι μια πολύ καλή απάντηση για του οργανωτέ των γεγονότων τη 19η και 20η Δεκεμβρίου. Το τελευταίο σημείο που ανέφερε επίση ο κύριο Φίλο ήταν το θέμα τη φιλελευθερωποίηση προξενικών θεωρήσεων. Δεν επαρκεί αυτό. Είναι καιρό πια να σταματήσουμε το τείχος, το χρηματοοικονομικό τείχος το οποίο έχει δημιουργηθεί για να προστατεύσει τον Λουκασέγκο και τους δικούς του μετά πριν από μερικά χρόνια. Ευχαριστώ κύριε Παλέσχης, ο κύριος Τζιγκέρης, ο οποίος είναι πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου της Λιθουανίας και που ε, έχει γίνει μια αντίστοιχη ακρόαση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μόλις προ λίγων ημερών οργανώσαμε ε, ακρόαση στο Λιθουανικό Κοινοβούλιο μετά από τα γεγονότα του Δεκεμβρίου στη Λευκορωσία και με συμμετοχή και του κ. Σουσκίεβιτς τα γεγονότα αυτά ξεπλούν κάθε φαντασία. Μας είπαν για παράδειγμα και ε, Νικλάγεβα μας είπε ότι έφεραν τον πατέρα της Μισόγυμνο οι άνθρωποι της ΚΑΚΕΜΠΕ και τον πήραν από το νοσοκομείο και τον πήγαν στη φυλακή. Στερούν οποιαδήποτε ιατρομοφαρμακευτική περίθαλψη από τους κρατουμένου. Ξεπερούν κάθε φαντασία. Φοιτητέ δικοί μα από τη Βίλνιους, Λευκορωσικό ε, Πανεπιστήμιο συνελήφθησαν. Μην ε, λησμονούμε ότι υπάρχουν και αγνοούμενοι και δεν υπάρχει και καμία ε, σοβαρή έρευνα για την τύχη τους. Πολιτικώς αντιφρονούντες δηλαδή. Χρειαζόμαστε λοιπόν πράγματι μια νέα στρατηγική. Συμφωνώ απόλυτα με τον Επίτροπο κύριο Φιούλε καθώς και με τις παρατηρήσεις του κύριου Γνατάγεβιτς αλλά οι νέες εκλογές που θα πρέπει να γίνουν. Θα πρέπει να γίνουν όντως στην Λευκορωσία. Θα πρέπει να προκυριχθούν νέες εκλογές καθώς και νέο συντονιστή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σχέση με τη Λευκορωσία. Και τον κατάλογο των κυρώσεων θα πρέπει να περιληφθούν και άλλα πρόσωπα που άσκησαν τρομοκρατική βία σε βάρος των αντιφρονούντων. Και πρέπει να δούμε και ποιες είναι οι σχέσεις που επηρεάζουν την εσωτερική κατάσταση στην Λευκορωσία. Και βέβαια το τελευταίο μου θέμα είναι θα πρέπει να ενισχύσουμε τις διακομματικές σχέσεις. Έχουμε εδώ κοντά μας τον κύριο Κασούριν, σοσιαλδημοκράτη, έχουμε εκπροσώπους από χριστιανοδημοκρατικά κόμματα, ορισμένοι βρίσκονται στις φυλακές, αλλά θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τα κοινοβουλευτικά μας κόμματα να συνεργαστούν με τα φύλλα κόμματα στη Λευκορωσία και να τους υποστηρίξουμε τώρα, ήδη τώρα. Νομίζω ότι όλα τα κόμματα τα παραδοσιακά κόμματα, είτε είναι το Λαϊκό Κόμμα, είτε το Σοσιαλιστικό, είτε άλλα αριστερά κόμματα, θα πρέπει να συνεργαστούν με τα αδελφά κόμματα στην ε, Λευκορωσία. Αύριο, 13 Ιανουαρίου, πριν από 20 χρόνια, ε, είχε γίνει, ε, είχαν γίνει παρόμοιες ταραχές στη Λιθουανία και εγώ γιορτάζουμε άλλωστε τώρα και τα 20 χρόνια από την πτώση του τείχους του Βερολίνου. Ακόμα έχουμε λοιπόν τώρα κρατούμενους στην ε, Λευκορωσία και εξακολουθούμε και έχουμε τείχος όχι πλέον του Βερολίνου αλλά στην, ε, μεταξύ ημών και της Λευκορωσίας. Ευχαριστώ κύριε Ζιγκέρης. Ο Σάιρος Βόλτς και έχει το λόγο. Ενάμιση λεπτό σε παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι προφανές το ότι πρέπει να καταδικάσουμε και να απαιτήσουμε, να εφαρμόσουμε κυρώσεις, ακόμα και να τις επεκτείνουμε και να εξετάσουμε την αναστολή της ε, εταιρικής σχέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ε, Λευκορωσία και τη συμμετοχή της στην ε, Euronest, όπως είχαν ζητήσει κάποιοι από την αρχή. Πρέπει να υποστηρίξουμε την κοινωνία των πολιτών, αλλά δεν αρκεί η ηθική υποστήριξη και οι καλές προθάσεις το πραγματικό γεωπολιτικό ερώτημα είναι κούι bono. Ποιο είναι αυτό ο οποίο κερδίζει από τα γεγονότα στη Λευκορωσία. Δεύτερον, τα γεγονότα αυτή τη στιγμή παίζουν το παιχνίδι τη Ρωσία. Τρίτον, τα γεγονότα αυξάνουν την απόσταση μεταξύ Λευκορωσία και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέταρτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Δύση αντιμετωπίζουν τα θέματα αυτά ω ο του Παύλοφ, όπω είπε και ο κύριο Στάνοκ βοηθούν ακριβώ αυτού που θέλουν μεγαλύτερη απόσταση Λευκορωσία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. σω το έχουν σχεδιάσει και έτσι. Τι πρέπει να κάνουμε στο μέλλον. Μία δίτη προσέγγιση χρειάζεται, όπω προτείνατε. Κυρώσει και απομόνωση τη κυβέρνηση, αλλά άνοιγμα προ την κοινωνία των πολιτών και μεγαλύτερη αρρωγή. Να ανοίξουμε την πόρτα τη Ευρώπη στη Λευκορωσία, αυτή είναι η καλύτερη κύρωση που μπορούμε να εφαρμόσουμε στο καθεστώ του Λουκασέγκο. Πρέπει να έχουμε μία μακρόπνοα στρατηγική για τα επόμενα δέκα χρόνια ο στρατηγικό μα εταίρο είναι η κοινωνία των πολιτών και όχι η κυβέρνηση. Ο στόχο μα είναι να προωθήσουμε τι ευρωπαϊκέ αρχέ και να προετοιμάσουμε νέε γενιέ Ευρωπαίων. Λένε μερικοί ότι είμαστε παγιδευμένοι μεταξύ τη αδιαφορία τη Αμερικανική κυβέρνηση, τη ανικανότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη πίεση τη Ρωσία στη Λευκορωσία. Έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση όμω όλα αυτά τα οποία έπρεπε να κάνει. Όχι. Ήμασταν διστακτικοί Πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Η Λευκορωσία είναι μια πραγματική δοκιμασία για τη νέα εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς το παρόν δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Λευκορωσία, οι Λευκορώσοι δημοκράτες οι οποίοι αποφασίζουν για τα γεγονότα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε υποχώρωση και από τη Λευκορωσία και από την Ουκρανία. Δεν πρέπει λοιπόν να το παραγνωρίσουμε αυτό και δεν πρέπει να αυτό ικανοποιούμεθα. Ευχαριστώ κύριε Σάιρους Βόλς και ο κύριος Σίρετς για μισή λεπτό. Ευχαριστώ. Είναι μια πολύ θετική ατμόσφαιρα, μια ωραία ατμόσφαιρα. Εμεί οι πολιτικοί αρεσκόμαστε στο να μιλάμε και αισθάνομαι πάντα πολύ καλά όταν βρίσκομαι σε μια τέτοια ρητορική ατμόσφαιρα. Αναρωτιέμαι όμως τι θα απογίνουν οι φιλοξενούμενοι μας όταν θα γυρίσουν πίσω στο Μίνσκ και θα πρέπει να μιλήσουν στους πολίτες τους να τους πούνε τι κάνανε εδώ που ήρθαν στις Βρυξέλλες, πόσα λεφτά τους δώσαμε παραπάνω για να πάνε στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, για να βοηθήσουν την ε, ε, πολιτική κοινωνία. Όλη αυτή ε, η χειρονομία για τις θεωρήσεις τι σημαίνει, σημαίνει ότι με λιγότερα λεφτά κάποιος θα παίρνει λιγότερο θα, θα παίρνει τη βίζα του οι κάτοικοι του Κιέβου, λέει ο μιλητής, θα καταλαβαίνουν γιατί θα πληρώνουν λιγότερα λεφτά για τις βίζες, οι οποίες δεν θα τους δίνονται. Θα μπορούσε λοιπόν η Κομισιόν να μας υποβάλει μια συγκεκριμένη πρόταση όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Μια ρεαλιστική πρόταση σε πραγματική γλώσσα, κατανοητή γλώσσα για να έχει πραγματική επαφή με τους λευκορώσους πολίτες και να είναι αυτή η απάντησή μας έναντι των συμβάντων και του δικτάτορα. Εγώ πίστευα ότι μπορούσαν να αλλάξουν τα πράγματα με τον δικτάτορα, αλλά τελικά είδαμε που καταλήξαμε. Και Δεδομένου ότι δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, εμείς και οι υπόλοιπες χώρες πρέπει να ανασύρουμε τα συμπεράσματά μας. Η κυρία Σρέντερ. Ευχαριστώ. Είμαι μέλος της Αντιπροσωπείας Κοινοβουλευτικών Σχέσεων Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Λευκορωσικού Κοινοβουλίου. Μέχρι τώρα δεν έχουμε κάνει κοινέ συνεδριάσεις. Εμείς το αποφασίσαμε αυτό. Δεν θέλουμε δηλαδή να υποστηρίξουμε δικτάτορες. Γνωρίζω την χώρα. Υπήρξα από το 1994 μέχρι το 2004 η συγκίτρια του Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό, για το θέμα της Λευκορωσίας. Είναι δηλαδή η περίοδος όπου εγκαθίδρυσε την εξουσία του ο Λουκασένκο. Έχουμε δει καταστάσεις που έχουν συμβεί και άλλοτε. Θυμούμε το 1997 όταν το Συμβούλιο Πολιτικών Εξωτερικών είχε εγκρίνει ένα σύντομο πρόγραμμα ανθρωπιστικής βοήθειας και υποστήριξης των δημοκρατικών δυνάμεων. Μέσα σε, μία, σε ένα μήνα επιτύχαμε να οδηγήσουμε το Συμβούλιο σε απόφαση και μάλιστα και για την χρηματοδότηση του προγράμματο. Ήταν πολύ δύσκολο βέβαια μετά να ιδρυθεί πράγματι ο μηχανισμό αυτό, αλλά επετεύχθη εν τέλει. Νομίζω παρόμοια μέτρα μπορούν να αποδείξουν την αξία του και να είναι επιτυχημένα. Όμω υπάρχουν και σημαντικότερα, πλεχιό πρόθεσμα μέτρα. Μέτρα τα οποία θα έχουν ανθρωπιστική βάση. Υπάρχουν κρατούμενοι που τώρα υφίστανται ποινικέ διώξει. πρέπει να του αναγνωρίσουμε ω πολιτικού κρατουμένου. Είναι πολύ σημαντικό σε κάθε δήλωση που γίνεται από μέρους μας αυτό να επαναλαμβάνεται ότι δεν είναι ποινική κρατούμενη, είναι πολιτική κρατούμενη. Έχουμε και ανθρωπιστικές καταστάσεις, οι οποίες αναφέρθηκαν προηγουμένως. Ένα μικρό παιδί δηλαδή, το οποίο αφαιρέθηκε από τους γονείς του. Και γνωρίζουν όσοι προέρχονται από την Ανατολική Γερμανία περί τίνος πρόκειται. Πρέπει λοιπόν να δραστηριοποιηθούμε άμεσα. Είναι από τα πιο σημαντικά μέτρα αυτά που μπορούμε να λάβουμε. Δεν μπορούν να συνεχιστούν αυτά τα πράγματα εκεί. Δεύτερο, η κατάσταση στη χώρα αυτή είναι τέτοια που ακόμα και οι συνήγοροι τώρα υφίστανται ποινικέ διώξει και κινδυνεύουν να χάσουν τι άδειε ασκήσεω επαγγέλματο. Και αυτά τα πράγματα πρέπει να λεχθούν λοιπόν. Στη στρατηγική μα θα πρέπει να υπάρξει και μια δεύτερη χρονική διάσταση. Αυτά όμως που σας είπα μόλις πρέπει να είναι τα πιο άμεσο πρόθεσμα μέτρα. Αντρικιένε 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ είμαι μέλος της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Λευκορωσία. Νομίζω ότι ήταν ένα σφάλμα να μην στείλουμε την Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία για την παρακολούθηση των εκλογών Έχουμε στείλει αντιπροσωπείε σε χώρε που είναι πολύ μακριά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή τη φορά δεν στείλαμε στον κοντινότερο γείτονά μα. Επίση, συμφωνώ ότι χρειάζεται μια διτή προσέγγιση. Κυρώσει εναντίον των υπευθύνων για την καταστολή και συγχρόνω πλήρη υποστήριξη, πλήρης υποστήριξη προ την αντιπολίτευση και του αγωνιστέ ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για του τελευταίου, κύριε Επίτροπε, δεν χρειάζεται να περιμένουμε τη συνδιάσκεψη των χορηγών ή οτιδήποτε τέτοιο. Πέρσι, όταν εγκρίθηκε, πέρσι εγκρίθηκε η έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε ήδη ένα κατάλογο μέτρων που προτείναμε. Φιλελευθερωποίηση για τις ε, ε, προξενικές θεωρήσεις. Σημεία επαφής για τις αντιπροσωπείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κτλ. Επίσης για τους νέους και τους φοιτητές, οι οποίοι βρίσκονται κάτω από μόνιμη απειλή. Έχουμε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Ανθρωπιστικών Θεμάτων στο Βίλνιους και ακόμα δεν έχουν καμία εγγύηση ότι θα τύχουν χρηματοδότηση φέτος και του χρόνου. Και αυτά συμβαίνουν σε μια τόσο κομβική και σημαντική στιγμή. Υπάρχουν τόσα πανεπιστήμια στην Ευρώπη που είναι έτοιμα να δεχτούν φοιτητέ από τη Λευκορωσία. Είναι καιρό να δράσουμε, να δράσουμε με συγκεκριμένο τρόπο και όχι μονάχα με ωραία λόγια. Ευχαριστώ κύριε Ο κύριος Μύρης και για μισή λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολλοί από εσά δεν έχετε πάει στη Λευκορωσία, ίσω εγώ όμω έχω πάει πολλέ φορέ, γνωρίζω πολύ καλά την κατάσταση και ξέρω ότι πραγματικά τα πράγματα είναι αποκαρδιωτικά. Και μέσα στα πλαίσια της τρέχουσας θητείας έχω πάει πολλές φορές στην Λευκορωσία για να δω την κατάσταση. Πρέπει να σκεφτούμε τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα και τι θα κάνουμε και στο μέλλον. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με, την, με τις επίσημες αρχές της Λευκορωσίας ή όχι. Ήμασταν αποτελεσματικοί στις δράσεις μας. Όχι, όχι και πάλι όχι. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση, γιατί όσο εμείς παραμένουμε στο επίπεδο ερωτήσεων και δεν δίνουμε απαντήσεις όπως τα ερωτήματα της συνεργασίας με τη Λευκορωσία στην Ευρωνάστ, ουσιαστικά εμείς δεν πρόκειται να αλλάξουμε με τον τρόπο αυτό την κατάσταση στη χώρα αυτή. Όταν δεν έχουμε καμία μακροπρόθεσμη στρατηγική ένα της Λευκορωσίας, δεν πρόκειται να αποκομίσουμε κανένα αποτέλεσμα από τις ενέργειές μας. Και ένα τελευταίο σημείο που θέλω να αντιμετωπίσω. Η δημοκρατία στη Λευκορωσία θα μπορέσει να γίνει πραγματική όταν πραγματικά αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα ως Ευρωπαϊκή Ένωση το θέμα της Λευκορωσίας και δεν παριοριστούμε σε φραστικές δηλώσεις, αλλά όταν περάσουμε στις πράξεις, ακόμα και συνεργασία με την κυβέρνηση της χώρας αυτής. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλες τις ευκαιρίες. Ευχαριστώ κύριε Μίλσκι. Ο κύριος Τόλκες για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι από τη Λευκορωσία. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε καταρχήν να εκφράσω την πλήρη συμπαράστασή μου προς εσάς και στην κυρία Νεβέτιεβα να εκφράσω την πλήρη συμπαράστασή μου και την υποστήριξή μου για τα γεγονότα της 19ης ε, Δεκεμβρίου και την κατάσταση του πατέρα σας που βρίσκεται τώρα στη φυλακή κάτω από εκτρές συνθήκες. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσφατα έχει πρόσφατα αποκηρύξει την ιδέα του να εξισωθούν τα αδικήματα του κομμουνισμού με τα αδικήματα του φασισμού και του ναζισμού την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Εμείς θα πρέπει να έχουμε μια πολύ πιο εύκαμπτη αντιμετώπιση έναντι του, της εποχής του κομμουνισμού από ό,τι στο παρελθόν. Βλέπουμε όμως τώρα τον Λουκασένκο, ο οποίος είναι ένας μετακομμουνιστικός δικτάτορας, και γνωρίζουν όλες οι χώρες της περιοχής, οι βαλτικές χώρες, η Ουγγαρία και η Ρουμανία ότι όλα αυτά είναι ουσιαστικά το κληροδότημα του κομμουνισμού και της κομμουνιστικής εποχής. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μια πιο στρατηγική σκέψη για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τις χώρες αυτές οι οποίες ε, είναι συνέχεια και αποτέλεσμα μιας κομμουνιστικής εποχής και πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε με ένα καλύτερο τρόπο τα προβλήματα των χωρών αυτό και κυρίως πώς θα πρέπει να δώσουμε μια μεγαλύτερη έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα και όχι να τα θυσιάσουμε στο, δωμό, στο βωμό των ε, οικονομικών συμφερόντων. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε λοιπόν στους ε, δικτάτορες να πάρουν τη σκητάλη από την κομμουνιστική ε, εποχή και παράδοση με τέτοιο τρόπο. Το τόνισε και ο Βίκτορ Ορμπαν στη χώρα μα και αυτό ισχύει και για χώρε όπω είναι η Σερβία. Δεν πρέπει λοιπόν να αφήσουμε αυτέ τι χώρε να εμποδίσουν την προσπάθεια δημοκρατία στην Ανατολική Ευρώπη. Η κυρία Γκόμε ε, θα κλείσει τη συζήτηση για ένα μισή λεπτά. Αυτό που διακρίνει ε, μια δικτατορία και ένα δικτάτορα δεν είναι αν είναι κομμουνιστές ή όχι, αλλά ότι καταπιέζει τις ελευθερίες και στην ουσία καταπιέζει τους λαούς. Εμείς οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι αποτύχαμε με την προηγούμενη ήπια προσέγγιση που θεωρήσαμε ότι μπορούμε να συνεννοηθούμε με τον δικτάτορα και να καταφέρουμε να υιοθετήσει μερικές πιο ελεύθερες πρακτικές. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε λοιπόν στο business as usual, ούτε επιτρέπεται να δεχθούμε να μας εκβιάζουν. Θα πρέπει οι στόχοι μας να είναι απόλυση των κρατουμένων, ελεύθερη λειτουργία των μέσων ενημέρωσης και επανάληψη των εκλογών. Βεβαίως χρειαζόμαστε μια στρατηγική για να υποστηρίξουμε τον κόσμο, τα ελεύθερα μέσα ενημέρωσης, τις οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών, τους φοιτητές. Να ενισχύσουμε τη δημοκρατική αντιπολίτευση, τα κόμματα που έχουν δημοκρατική ατζέντα και βεβαίως να είμαστε πολύ αυστηροί σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις που θα επιβληθούν στο καθεστώς. Απαγόρευση ε, ταξιδιού, πάγωμα περιουσιακών του στοιχείων και εάν χρειαστεί και αναστολή της συμμετοχής τους στην ε, ε, πρωτοβουλία ε, Ανατολικής, γειτο... Ανατολικής Γειτονίας. Ο Πρόεδρος για την Επιτροπή των Σχέσεων με τη Λευκορωσία έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι περιορισμένος ο χρόνος και γι' αυτό δεν μπορέσαν καν όλοι οι προσκεκλημένοι μας από τη Λευκορωσία να λάβουν το λόγο έχουμε εδώ και τον κύριο Μιλίνκεβιτς αλλά και άλλους που μίλησαν όπως ο εκπρόσωπος των ελεύθερων δημοσιογράφων έχουμε όμως και τον κύριο Σουσκίεβιτς τον πρώην πολιτικό κρατούμενο δόκτωρα Αλεξάνδρ Καζόλιν τον επικεφαλής του εσωτερικού παρατηρίου, παρατηρητηρίου δημοκρατικών ε, αλλαγών αχ, συγγνώμη ξέχασα το όνομά του τον κύριο Γκαλιάκιν, λοιπόν πολύ και θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε βαθύτερα το θέμα αυτό στις 5 στην αίθουσα 3Ε2 με όλους τους λευκορώσους ε, προσκεκριμένους μας θα έχουμε και τη δυνατότητα να δούμε και κινητές εικόνες, να δούμε και ε, προβολή ταινίας με το τι συνέβη στο Μίνσκ στι 19 ε, και 20 Δεκεμβρίου. Αυτά ήθελα μόνο να πω. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Συμπεράσματα του κυρίου Μπούζεκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Για μας όλους το πιο σημαντικό στοιχείο ήταν οι συμβουλές που πήραμε από τους φίλους μας από τη Λευκορωσία. Μία άκαμπτη, μονοκόμματη ε, αντιμετώπιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πολιτική πίεση για τη χωρίς όρους απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων, όπως είπε η κυρία Νικλάγεβα, αυτό είναι το κλειδί στη φυλακή του πατέρα της. Πρέπει να εξασφαλίσουμε την πρόσβαση στην πληροφορία και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω να σας ευχαριστήσω λοιπόν όλους για τις απόψεις και τις γνώμες που συνεισφέρατε στη σημερινή συζήτηση. Μερικές σύντομες παρατηρήσεις που νομίζω ότι μπορούν να αποτελέσουν ένα πυρήνα συνένεσης για όλους και που προερχόνται και από την πρωινή μου συναντήση με όλους τους εκπροσώπους της λευκορωσικής αντιπολίτευσης. Διευκόνηση ε, προξενικών θεωρήσεων, διτή προσέγγιση, ελευθερία για τους πολίτες και ακόμα και κατάργηση για ορισμένε ομάδες ε, πολιτών όπως είναι οι φοιτητέ, οι καλλιτέχνες, οι επιστήμονες ενώ παράλληλα και ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρξει απαγόρευση ταξιδίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για όλους τους αξιωματούχου της Λευκορωσία που ενέχονται στα γεγονότα της 19 η 20 η Δεκεμβρίου. Η υποστήριξη για τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις τη κοινωνίας των πολιτών και φυσικά μεγαλύτερη χρηματοοικονομική υποστήριξη. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να βρούμε τρόπου, να υποστηρίξουμε τι ανεξάρτητες ΜΚΟ που αυτή τη στιγμή δεν έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στα μητρώα της Λευκορωσίας λόγω του αυταρχικού καθεστώτος της χώρας αυτής. Και φυσικά η υποστήριξη για τους φοιτητές και για τα πανεπιστήμια είναι πολύ σημαντική, χρηματική βοήθεια. Οι υποτροφίες θα πρέπει όλα αυτά να αυξηθούν και θα πρέπει να δώσουμε ένα καλό παράδειγμα όπως με το Πανεπιστήμιο του Βίλνιους για τις ανθρωπιστικές σπουδές που πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχουν και άλλε προτάσει τι οποίε θα πρέπει να σκεφτούμε Παραδείγματο χάρη, η έκκληση για την επανάληψη των εκλογών, όπω τόνισε ο κύριο Στάνο, και επίση έχουμε μία ακόμα πρόταση, η οποία δεν προέρχεται από αυτή τη συνεδρίαση, να μην συμμετάσχει η Λευκορωσία σε διεθνεί αθλητικού αγώνε, όπω είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνε και το Παγκόσμιο Κύπελο ε, Ποδοσφαίρου. Όσο δυνατό και να είναι. Αλλά υπάρχουν και άλλε προτάσει. Δεν πρέπει να σκεφτούμε για όλες αυτές τις προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να δούμε ποια θα πρέπει να είναι τα επόμενα βήματα που θα κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αύριο θα έχουμε συνέλευση των πρόεδρων των πολιτικών κομμάτων και θα ληφθεί μια απόφαση για την αποστολή μιας αντιπροσωπείας μιας εξεταστικής επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Λευκορωσία και επίσης θα υπάρξει συζήτηση κατεπηγόντων την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο και ψήφισμα για τη Λευκορωσία και στη συνέχεια εμείς θα πρέπει να αποφασίσουμε σε σχέση με τη συνέχιση ή αναστολή της συνεργασίας μας με τη Λευκορωσία μέσα στην Euronest. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν πρέπει να ληφθεί αυτή η απόφαση γιατί ήδη <clears throat> έχουμε περιμείνει ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και τώρα επιτέλους θα πρέπει να αποφασίσουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Και περιμένουμε επίσης και το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις 31 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες, που είναι πολύ σημαντικό και προσδοκούμε ότι θα υπάρξει και συνεχής επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Τέλος, θέλω να πω, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι, σήμερα υποδεχτήκαμε τους νικητές των εκλογών στη Λευκορωσία όχι επίσημα, αλλά από πολιτική και ψυχολογική άποψη αυτό κάναμε. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό εγχείρημα και τα πιο σημαντικά νέα από εμά. Και σας αντιμετωπίζουμε, φίλοι μας από τη Λευκορωσία, σαν νικητές των εκλογών και είμαστε σίγουροι ότι θα νικήσετε στις επόμενες εκλογές και σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε Μπούζεκ. Ευχαριστώ και τους λευκορώσους φίλους μας που συμμετείχαν δυναμικά στη συνάντηση και όλους τους συναδέλφους που μίλησαν. Πριν ολοκληρώσουμε τις εργασίες μας θα ήθελα να σας πω ότι οι πρόεδροι που κάθονται γύρω από αυτό το τραπέζι έχουν ετοιμάσει ένα κείμενο και μία δήλωση που θα ήθελα να σας παρουσιάσω σύντομα και που αποτελεί τα την περίληψη των συμπερασμάτων των όσων ακούστηκαν σήμερα. Πρόκειται για μια κοινή δήλωση γύρω από τα όσα συζητήσαμε, δηλαδή ότι οι εκλογές δεν ήταν ελεύθερες και δημοκρατικές σύμφωνα με τις διεθνείς ε, προδιαγραφές καταδικάζουμε την καταστολή των ειρηνικών διαδηλώσεων με τη βία με φυλακίσεις, κρατήσεις ε, και άλλα επεισόδια Επίσης ε, καλούμε σε γενική σκέψη γύρω από τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις αρχές της Λευκορωσίας. Καλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να απαγορεύσει τη χορήγηση θεώρηση σε όλους τους ε, αξιωματούχους οι οποίοι πήραν μέρος ε, στην καταστολή των διαδηλώσεων. Ζητούμε την άμεση απολευθέρωση των προσωπικότητων που κρατούνται η χρηματική ενίσχυση των ανεξαρτήτων ΜΜΕ, των μη κυβερνητικών οργανώσεων, της κοινωνίας, δηλαδή των πολιτών της ε, Λευκορωσίας, των οργανώσεων εκείνων που ασχολούνται με την ε, ενίσχυση της ε, δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ζητάμε την αύξηση των υποτροφιών για τους Λευκορώσους φοιτητές ε, ζητούμε τη μείωση του κόστου των θεωρήσεων για τους φοιτητές, τους επιστήμονες, τους καλλιτέχνες. ενίσχυση των διακοινοβουλευτικών μας σχέσεων με τη Λευκορωσία στα πλαίσια της Euronest και τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό ζητούμε από τις λευκορωσικές αρχές να αναστείλουν την απαγόρευση λειτουργίας του γραφείου της ΟΑΣΕ στο Μίνσκ. Ελπίζω ότι έτσι τα βλέπετε κι εσείς και καλύπτουμε δηλαδή την σκέψη σας αλλά και τον προβληματισμό της ε, λευκορωσικής ε, κοινωνίας. Σας ευχαριστώ όλους και εύχομαι να ξανασυναντηθούμε σύντομα με μια βελτιωμένη κατάσταση όπως όλοι ευχόμαστε.